Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, θα ήθελα να ξεκινήσουμε, αν γίνεται. Έχετε λάβει καιρος την, το σχέδιο μέρησης διάταξης και θα σας πρότεινα να την ακολουθήσουμε. Καταρχήν το πρώτο σημείο, έγκριση. Υπάρχουν μήπω παρατηρήσει αντιρρήσει ω προ το σχέδιο τη διάταξη που σα στείλαμε. Όχι, πολύ ωραία, οπότε εγκρίνεται. Έχω κάποιε ανακοινώσει πριν περάσουμε στη, στα ουσιαστικά θέματα ε, με του καλεσμένου μας. Ανακοινώσει. Καταρχήν, συνεδρίαση τη 15 η Μαρτίου. Οι συντονιστές ε, συμφώνησαν ω προ τη Στρογγυλή Τράπεζα για την ανάγκη διεθνού συνεργασίας ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα των θυμάτων της Τρομοκρατία και μάλιστα αυτό θα γίνει σε συνεργασία με τις Επιτροπές ΛΥΜΠΕ και ε, ΔΡΟΑ όπως ενέκριναν οι συντονιστέ και θα γίνει στις 24 Μαΐου 3 με 5 στα πλαίσια της συνεδρίαση τη Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών τη ΛΥΜΠΕ. Δεύτερη ανακοίνωση. Η αποστολή της Επιτροπής μας στη Μαδρίτη θα λάβει χώρα 9 με 11 Μαΐου τρέχοντος έτους. Ανακοίνωση τρίτη. Η αποστολή της Επιτροπής μας στην Κατάνια με μία, μισή μία μέρα στη Ρώμη θα γίνει 6 με 8 Ιουνίου του 2018 όπως αποφάσισαν οι συντονιστές και τέταρτη και τελευταία ανακοίνωση ο Επίτροπος Έτιγκερ θα προσκληθεί σε μια μελλοντική συνεδρίαση της Επιτροπής μας για να μας μιλήσει για τους υπάρχοντες πόρους ό,τι αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Γιατί αυτό είναι και ένα από τα θέματα της εντολής της Επιτροπής, της Επιτροπής ΤΕΡ της δικής μας. Αυτά ως προς ανακοινώσεις και θα πρότεινα τώρα να υποδεχθούμε τον κύριο Ζανσάλ Μπριζάρ, τον πρόεδρο του Κέντρου Ανάλυσης της Τρομοκρατίας, του ΚΑΤ δηλαδή, στη Γαλλία. Ζητήσαμε να έρθει να μας μιλήσει και να συζητήσουμε μαζί του, γιατί όχι μόνο έχει τεράστια αναλυτική και αναγνωρισμένη και φημισμένη αναλυτική ικανότητα, αλλά και λόγω της προσωπικής του πορείας ο κύριος Πριζάρα ε, έγινε κατεξοχήν συνομιλητής ε, ε, της Επιτροπής μας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και μάλιστα μετά τις νομικές σπουδές που έκανε στη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία σε επαφή με τα μυστήρια της εξουσίας και τους μοιημένους εξουσίας στη Γαλλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, καταρχήν ήταν ε, στο προσωπικό γραφείο του Πρωθυπουργού Εντουάρ Μπαλαντούρ, μετά ήταν συνεργάτης ε, ε κοινοβουλευτικό στην Εθνοσυνέλευση και κατόπιν συνεργάστηκε με τον ε, δικαστή Αλέ Μαρσό, ε, υπεύθυνο της αντιτρομοκρατικής μονάδας στο Παρίσι. Κατόπιν ανέλαβε θέματα ασφάλειας και πληροφοριών οικονομικών και στα τέλη του προηγούμενου αιώνα, μου αρέσει να το λέω έτσι, δηλαδή γύρω στο 1999, ε, ειδικεύεται στην κρυπτογράφηση των κυκλωμάτων χρηματοδότησης των μουσουλμανικών και κυβερνητικών οργανώσεων ε, ε, που είχαν διασυνδέσει με το κίνημα των ριζοσπαστικών Ισλαμιστών. Και μάλιστα η έκθεσή του μετονομάστηκε μετά τις επιθέσεις του 11 Σεπτεμβρίου 2001 έκθεση για το οικονομικό περιβάλλον του Σάμα Μπεν Λαντέν. Μάλιστα, είχε μεγάλη απήχηση στα ΜΜΕ. Και μετά, μάλιστα, από συνεργασία του με πολλές επιχειρήσεις, ε, ασχολήθηκε με θέματα οικονομικής, οικονομικών πληροφοριών, διεθνούς ε, ε, δικαίου και θέματα επικοινωνίας και θέματα κρίσεων. Μάλιστα, κάνει συχνέ παρεμβάσει στα ΜΜΕ λόγω των μεγάλων των γνώσεων για την τρομοκρατία και τη χρηματοδότησή τη. Και μάλιστα το Κέντρο Ανάλυση Τρομοκρατία, στο οποίο προεδρεύει, δημοσίευσε στι 23 Φεβρουαρίου, παρελθόντος Φεβρουαρίου, μια έκθεση με τίτλο «Η τρομοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Άνω και κάτω τελεία, απολογισμό του 2017. Και μάλιστα η έκθεση αυτή κάνει έναν γενικό απολογισμό, μια επισκόπηση ε, του θέματος αυτού και μια επικαιροποίηση ε, που είναι πολύ ευπρόσδεκτη και στα πλαίσια των δικών μας εργασιών. Θα μας τα πει αυτά αργότερα. Θα του πρότεινα λοιπόν να μας παρουσιάσει τον απολογισμό του 2017 όπως φαίνεται στην έκθεση του ΚΑΤ και μετά θα γίνει συζήτηση όπου οι συνάδελφοι θα παρουσιάσουν τις απορίες του και φαντάζομαι θα λυθούν ε, χάρη στον καλεσμένο μας ε, για τα θέματα χρηματοδότηση τη τρομοκρατία. Χωρί άλλη χρονοτριβή, λοιπόν, κύριε Μπριζάρ, σα δίνω το λόγο για ένα 20 λεπτό περίπου, αν δεν έχετε αντίρρηση φυσικά. Είπατε προηγουμένω ότι συμφωνείτε. Και κατόπιν ο κύριο Μπριζάρ συμφώνησε να ακολουθήσουμε τη δική μα μέθοδο του πινκ-πονγκ, δηλαδή να δίνουμε το λόγο σε κάθε μέλος για να υποβάλει τι ερωτήσει του και αμέσω στον καλεσμένο μα για να δίνει απαντήσει. Αυτά και έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καταρχήν, να κάνω μια επισκόπηση της κατάστασης και της απειλής τη τρομοκρατικής στην Ευρώπη κυρίως, πριν περάσω στις νέες προκλήσεις σε αυτή την προσπάθεια καταπολέμησης τρομοκρατίας με τον τρόπο που έχει αναδιαμορφωθεί και η τρομοκρατική απειλή. Καταρχήν, έχουμε μια υποχώρηση εδαφική του Ισλαμικού κράτου στη Συρία και το Ιράκ, που δεν μείωσε όμω μηχανικά το επίπεδο τη απειλή. Και ναι, βέβαια, επηρέασε τι επιχειρησιακέ ικανότητε τη οργάνωση αυτή και αποδιοργάνωσε τη, το προπαγανδιστικό του σύστημα, παρόλα αυτά δεν το εκμηδένισε. Και μάλιστα στην τελευταία μελέτη του Κέντρου Ανάλυση Τρομοκρατία για την επισκόπηση τη τρομοκρατία το 2017, είδαμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πέρυσι είχαμε 62 τέτοια ε, τρομοκρατικά επεισόδια που έχουν σχέση με τη σφαιρολογική σύνδραση. Ε, σύγκρουση 15 μάλιστα από αυτά ε, διαπράχθηκαν 40 καταφέραμε να τα αποτρέψουμε και μάλιστα τα περισσότερα, τα μισά μάλλον έγιναν στη Γαλλία που είναι η πρώτη χώρα μετά το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία. Και από το 2013 η πατρίδα μου, η Γαλλία, ε, γνώρισε πολύ έντονη τρομοκρατική δραστηριότητα από όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, με το μισό, επαναλαμβάνω, των περιστατικών και των τρομοκρατικών επιθέσεων να γίνονται στο έδαφο τη. Και μάλιστα είχαμε μεγάλε τα 62 άτομα ε, νεκρού και πάνω από 200 τραυματίε. Και μάλιστα ε, ήταν το υψηλότερο ποσό του 2007. Τι διδαχθήκαμε από την έκθεση αυτή. Καταρχήν, δεν έχει μειωθεί η ένταση αυτή τη απειλή παρά την υποχώρηση του Ισλαμικού κράτους στην εδαφική. Επίσης, είχαμε μείωση ε, των, της αποχώρησης των ε, ξένων μαχητών, αλλά έχουμε παρουσία σημαντική. Το 45% των ε, επιθέσεων αφορούσαν αστυνομικέ και στρατιωτικέ δυνάμεις και το υπόλοιπο ποσοστό ήταν κατά αμάχων. Επίσης, ένα τρίτο των ε, όπλων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ε, ε, ε κυρίως μαχαίρια, ε, λευκά όπλα, κάτι που δείχνει την ε, αποτελεσματικότητα που έχουν ε, τα εγχειρίδια για την παρασκευή και αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών που κυκλοφορούν στο διαδικτύο. Άλλο που διδαχθήκαμε πάνω από το 50% των δραστών των τρομοκρατικών επιθέσεων στην Ευρώπη ήταν, από τη... ήταν υπήκοοι της χώρας στην οποία έδρασαν και 10% αυτών είχαν πραγματοποιήσει παραμονή στη, στο Συρία-Ιράκ. 10% δηλαδή αυτών είχαν επιστρέψει. 50% ήταν άγνωστοι δράστες στις, μονα, στις υπηρεσίες, στις μυστικές, τη στιγμή που δραστηριοποιήθηκαν. Κάτι που δείχνει ακριβώς το εύρος της απειλής. Άλλο ε, δίδαγμα σε ό,τι αφορά τη σχέση των δραστών και των τρομοκρατικών οργανώσεων. 47% των επιθέσεων εμπνεύστηκαν χωρίς να έχουν άμεσο, άμεσο σύνδεσμο με τις τρομοκρατικές οργανώσεις. 45-47%. Ε, ένα μεγάλο ποσοστό ήταν τηλεκατευθυνόμενο από άτομα που στη χώρα προέλευσης είχαν κάποια σχέση με τζιχαντιστές που δραστηριοποιούνταν επιτόπου και 8% ήταν ε, κατευθυνόμενες ε, από ε, επιστρέφοντες ξένους μαχητές και που είχαν εκπαιδευτεί στις εμπόλεμες περιοχές και επιστρέψει στην Ευρώπη για να χτυπήσουν. Αυτό που δείχνει τελικά η μελέτη και αυτό που παρατηρούμε μετά από αυτή την κατεπίγουσα κλίση που ακούω, αυτό που παρατηρούμε λοιπόν είναι ότι οι προβλεπόμενη εξαφάνιση του Ισλαμικού κράτου δεν θα οδηγήσει σε εξαφάνιση τη τρομοκρατική απειλή, Για δύο λόγου κυρίως. Γιατί οι βασικοί φορεί της τρομοκρατική απειλή σήμερα, η καιντα και το Ισλαμικό κράτος, έχουν αποδείξει την ανθεκτικότητά του. Το 2009 οι Αμερικανοί έλεγαν για τον προκάτοχο του Ισλαμικού κράτου ότι ε, είχε ξεριζωθεί πλήρω είχε εξαλειφθεί. Επίσης αυτές οι δύο οργανώσεις έχουν ε, χιλιάδες παρακλάδια ανά τον κόσμο που εξασφαλίζουν τη μακροβιότητα της τρομοκρατικής απειλής. Και μπορεί η Αλκάιδα να έχασε στο Αφγανιστάν ε, μεγάλο έδαφος, ε, αλλά το Ισλαμικό κράτος αντίθετα μετατράπηκε από τρομοκρατική ομάδα σε τρομοκρατικό δίκτυο. Αντίθετα από την Αλκάιδα που είχε αντίστροφη πορεία. Και έχουμε μια παγκοσμιοποίηση του Ισλαμικού κράτου. Ουσιαστικά. Επίση από τον Νοέμβριο του 2017 ο ηγέτης του Ισλαμικού κράτους κάλεσε όσους δεν μπορούσαν να έρθουν στην καρδιά του χαλιφάτου να πάνε σε άλλες επαρχίες του Ισλαμικού κράτους και να δραστηριοποιηθούν. Και μάλιστα ξέρουμε ότι δραστηριοποιήθηκα στην Αφρική, την Ιεμένη, το Αφγανιστάν, στην Νοτιοανατολική Ασία. Και επίσης είχαμε ε, πολλούς πυρήνες τρομοκρατικούς και στην Ευρώπη, όπως είδαμε από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες. Επίσης, ε, ως ό,τι αφορά τους ξένους μαχητές που στρατολογήθηκαν ε, από το Ισλαμικό κράτος στη Συρία και το Ιράκ και κατόπιν ε, ε, μετέβησαν στο Αφγανιστάν ή στη Λιβύη. Κατέχουμε τέτοιες πληροφορίες. Επίσης, τα παρακλάδια έχουν αναπτύξει και δράση εκτός του, της επικράτειας του Ισλαμικού κράτους. Το 2016 ε, το παρακλάδι του Ισλαμικού κράτους στο Αφγανιστάν έχει ε, σχέση με, ένα, τρομοκρατική επίθεση στη Νέα Υόρκη. Επίσης ε, στο Μάντσεστερ μια επίθεση είχε διασυνδέσεις με αντίστοιχα παρακλάδια. Επίσης μια, ένα παρακλάδι της Αλκάιντα, το Αλκπα, έλαβε το σκητάλι από την κεντρική Αλκάιντα μετά την υποχώρηση που παρουσίασε στο Αφγανιστάν και μάλιστα η ΑΚΠΑ από το 2009 πολλαπλασίασε τα σχέδια τρομοκρατικών επιθέσεων και αποπειρών στις δυτικές χώρες, αναπτύσσοντας μια αυτόνομη ικανότητα ε, προπαγάνδας και ε, επιχειρησιακής δραστηριότητας. Οπότε έχουμε μια ε, μετεγκατάσταση αυτής της επιχειρησιακής δραστηριότητας σε εδάφη μακριά από το Ισλαμικό κράτος. Αυτό παρατηρούμε σήμερα και μάλιστα ε, τέτοιες δραστηριότητες στηρίζονται οικονομικά και από το Ισλαμικό κράτος, από την Κεντρική Επιτροπή, γιατί διαπιστώνουμε μεταφορά ε, χρημάτων από, την, ε, από το Ιράκ προς τα παρακλάδια του Αφγανιστάν, της Ιεμένης και της Νοτιοανατολικής Ασίας. Επίσης, ε, διαπιστώνουμε την επιθυμία των ξένων μαχητών όχι να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, ε, στη χώρα προέλευσης, αλλά να μεταβούν σε άλλους θύλακες που ελέγχονται από το Ισλαμικό κράτος στη Συρία και το Ιράκ ή σε ε, παραμεθόριες χώρες πριν μετακαταστούν σε άλλες εμπόλεμες ζώνες, τη Λιβύη, το Αφγανιστάν, τη Λιβύη, το Αφγανιστάν Μαλαισία και ούτω καθεξής. Έχουμε ακόμη την, τις αποδείξεις ότι μαχικές από το Ιράκ και τη Συρία έχουν μεταναστεύσει προς τη Λιβύη ή το Αφγανιστάν. Οπότε εξωγενείς απειλές για το, κατά το μοντέλο των τρομοκρατικών επιθέσεων του Βασίου και των Βρυξελών υπάρχουν ακόμη. Παρόλο που το Ισλαμικό κράτος παρεμποδίζεται στη δράση του στην στον πυρήνα του στο, στη Συρία και το Ιράκ. Επίσης, ε, έχουμε παρατηρήσει μια ανασύνθεση των, των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων μέσω της ενίσχυσης των παρακλαδιών, των θηγατρικών κατά κάποιο τρόπο του Ισλαμικού κράτους. Επίσης, έχουμε ένα κατακαιρματισμό της τρομοκρατικής απειλής, μια παγκοσμιοποίηση, όπως σας είπα, της απειλής. Ε, όπως παρατηρήσαμε και με τη, με τη βάση της Αλκάιντα. Ε, η τρομοκρατική απειλή διαιωνίζεται γιατί το Ισλαμικό κράτο και άλλε τρομοκρατικέ οργανώσει καταφέρουν να κινητοποιήσουν τους οπαδού του και να εμπνεύσουν άλλους. Και μπορεί μετά την εδαφική ήττα να μειώθηκε κάπως το Ισλαμικό κράτος και παρόλα αυτά διαπιστώνουμε ότι δεν καταφέραμε να οριοθετήσουμε ή να περιορίσουμε την απειλή. Και το να μειώσουμε το, το Ισλαμικό κράτος εδαφικά θεωρώντας ότι η τρομοκρατική απειλή θα περιοριστεί δεν είναι σωστό. Γιατί το Ισλαμικό κράτος δεν έχει μόνο εδαφικές βλέψεις. Γιατί πολλοί το 2014 θεώρησαν ότι το Ισλαμικό κράτος δεν πρόκειται να στραφεί, να επιτεθεί σε δυτικές οργανώσεις, ότι είχε μόνο εδαφικές βλέψεις και περιφερειακές. Αυτό όμως διαψεύστηκε. Και σίγουρα υπάρχουν και ενδογενεί λόγια τη απειλή. Ε, υπάρχει τηλεκατεύθυνση από εξωτερικέ ζώνε ή έμπνευση από την δρομοκρατική προπαγάνδα. Η απειλή είναι διάχυτη ε, και δεν υπάρχει χαρακτηριστικό προφίλ των δραστών. Ε, η, τα όπλα μερικές φορές είναι αυτοσχέδια και δεν υπάρχει και μια κοινή λογική, δεν υπάρχει ένα μύθος αριάδενης Επίσης, ε, ο δεσμός μεταξύ των δραστών και των δημοκρατικών οργανώσεων είναι όλο και πιο εικονικός. Και μάλιστα αυτός ο ενδογενής αυτή η ερασιτεχνική τρομοκρατία δεν είναι καινούρια. Και άλλες οργανώσεις πριν από το, το κράτος είχε, πριν από το Ισλαμικό κράτος είχαν δοκιμαστεί. Και μάλιστα το Ισλαμικό κράτος έχει αναφεράγει λογικές που προϋπήρχαν με τη διαφορά ότι το μήνυμά του πια έχει μαζική διάδοση και η δυνατότητα κινητοποίησης είναι τεράστια. Σε μεγάλο βαθμό λοιπόν το Ισλαμικό κράτος είναι η προέκταση κατά κάποιο τρόπο του, της Αλκάιντα, ενώ έχει άλλα μέσα και άλλες φιλοδοξίες από την Αλκάιντα. Γιατί η διατήρηση της απειλής οφείλεται και στους δράστες αυτής της ε, ιδεολογίας. Το εικονικό αυτό χαλιφάτο που θέλει να, να αυξήσει τους οπαδούς και να δώσει ε, συμβουλές μέσω χειριδίων κατασκευής εκρηκτικών μηχανισμών. Και μάλιστα αυτός ο παράγοντας ε, τε, ουσιαστικά γαλουχείται από την ριζοσπαστικοποίηση, τρέφεται από αυτή και προσαρμόζεται στις στους περιορισμούς ασφαλείας ε, που επιβάλλονται από τις ε, κάστε κοινωνίες. Τώρα, ποιες είναι οι προκλήσεις αυτής της κατάστασης και πώς ε, μετατρέπεται, μεταμορφώνεται σταδιακά η τρομοκρατική απειλή. Καταρχήν, ριζοσπαστικοποίηση. Αυτό αποτελεί ένα βασικό διακύβευμα, γιατί αυτό θα μας απασχολήσει για πάρα πολλά χρόνια και επίσης 50.000-60.000 ε, ε, είναι τα άτομα στην Ευρώπη τα οποία θεωρούμε ότι είναι ρίζους παστικοποιημένα σε διάφορες μεγάλες χώρες. 20.000 δηλαδή τέτοια άτομα στην Γαλλία και μόνο. Και να σας υπενθυμίσω και δύο άλλα στοιχεία. 60% αυτών που έχουν πληχτεί που μας έχουν πλήξει μάλλον ε, στην Γαλλία από το 2013 και μετά είναι άγνωστοι, δεν έχουν στοιχεία στις στη Γαλλική αστυνομία και πάνω από 50% των καταδικασμών για τρομοκρατικέ πράξεις από το 2014 είχαν α, ε, ε, λευκό ποινικό, μητρό. Δεν είχαν δηλαδή, δεν ήταν γνωστοί στην αστυνομία. Σε ό,τι αφορά τώρα την προληπτική δράση και εξουβετέρωση, σε ό,τι αφορά και τι μυστικέ υπηρεσίε. αυτό φυσικά είναι δική τους αρμοδιότητα και Πρέπει να πούμε ότι η μαζική αυτή διάσταση της ιστορικής απειλής σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει κινητοποίηση όλων των φορέων και των τοπικών αλλά και όλων των υπόλοιπων φορέων που πλήττονται από την ε, τρομοκρατία. Το μοντέλο από το 1986 στην Ευρώπη και στην Γαλλία ήταν ε, η κεντρική διαμόρφωση και εξειδίκευση της ε, προληπτικής και αποτρεπτικής ε, αντιμετώπισης της τρομοκρατίας και κυρίως της ομαδικής τρομοκρατίας κατά του κράτους. Και το σύστημα αυτό όμως έχει πλέον, είναι παροχημένο πλέον γιατί δεν υπάρχουν ίδιες απειλές σε ό,τι αφορά για παράδειγμα το τοπικό τους χαρακτήρα και η απειλή είναι πανταχού παρούσα και δεν ε, μπορεί πάντα δυστυχώς να εντοπίζεται. Άρα ο ρόλος ε, των τοπικών φορέων, των ε, δημάρχων, των τοπικών φορέων είναι πραγματικά κρίσιμος. Γιατί είναι αυτή στην πρώτη γραμμή σε ό,τι αφορά την εντοπισμό των φαινομένων, των συμπτωμάτων ριζοσπαστικοποίησης, γιατί προφανώς υπάρχει και κοινωνική και εκπαιδευτική διάσταση και σε ό,τι αφορά προφανώς και την ασφάλεια των κοινών χώρων και του ε, κοινού, του κόσμου. Και αυτό προφανώς σημαίνει μια διαφορετική πραγματικότητα και μια διαφορετική διάδραση, διάδραση που χρειάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την ασφάλεια των πόλεων υπάρχουν νέα μοντέλα. Δεύτερο διακύβευμα αυτό το θέμα των επιστροφών. Οι επιστροφές αυτές ε, νομίζω ότι έχουν προκαλέσει μεγάλους ε, φόβους. Τι διαπιστάνουμε λοιπόν σήμερα. Διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει μαζική ε, επιστροφή σε τόπους που έχουν επλεχθεί από τραποκρατικά κρούσματα στο 2017 ή στη Γαλλία έχουν καταγραφεί 14 επιστροφές. επιστροφέ. Οι μητέρε ήταν γυναίκε και παιδιά. Στο Βέλγιο και στη Γερμανία λιγότερε από 10 τέτοιε επιστροφέ. Και έτσι λοιπόν Υπάρχει μια τέτοια τάση πραγματικά. Οι άλλοι τζιχαντιστές ε, που θα συλληφθούν για παράδειγμα σε ε, ομάδες από το Ιράκ, από τη Συρία και περνάνε δίκη από τις τοπικές αρχές. Και θα πρέπει να σας πενθυμίσω και κάποια σημεία στο σημείο αυτό, κάποια νομικά στοιχεία. Καταρχάς δεν υπάρχει οποιαδήποτε ε, διεθνής υποχρέωση για τις χώρες ε, να παίρνουν από δίκη όσους έχουν τους υπηκόους τους που έχουν διαπράξει τρομοκρατικές πράξεις. Και η συνθήκη της Γενέβης ε, σας ε, υπενθυμίσω ότι ισχύουν σε ό,τι αφορά διεθνείς συγκρούσεις, αναπλές συγκρούσεις. Δίνουν ε, αρμοδιότητα στις ένοπλες ομάδες να κρίνουν αυτούς που να παίρνουν αποδίκη, αυτού που, που προβαίνουν σε επιθέσεις. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τον επαναπατρισμό των ε, υπευθύνων και σε ό,τι αφορά την δυνατότητα να ζητήσουν ε, αμνηστία από τις ε, τοπικές αρχές. Άρα, οι επιστροφές αυτές παραδόξως εκπροσωπούν πιο πολύ μια εξωτερική απειλή και όχι τόσο μια εσωτερική απειλή σε βραχυπροθεσμό και μεσοπροθεσμό επίπεδο. Και να μην ξεχνάμε και την, ε, τις περιπτώσεις των ε, Αφγανών, για παράδειγμα, που έκαναν επιθέσεις. Ε, θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη ανταλλαγή απόψεων πληροφοριών και καλύτερη συνεργασία με τρεις, χώρ, χώρες σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση των τζιχαντιστών. Ένα άλλο θέμα σε ό,τι αφορά την επιστροφή αφορά αυτούς που έχουν ήδη μπει, για παράδειγμα, στη Γαλλία. Για παράδειγμα, 70, έχουμε, στην Γαλλία έχουμε 258 ενήλικες που έχουν επιστρέψει το 2012. 76 αυτών είναι σε κράτηση και περιμένουν την δίκη τους. Και 64% αυτών θα έχουν ολοκληρώσει την, ε, κατά την ποινές μέχρι το 2020. Άρα ε, το μέσος όρος της ποινή είναι περίπου 7 χρόνια φυλάκιση. Και έτσι λοιπόν ε, γι' αυτό καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι 64% θα έχουν απελευθερωθεί πριν από το 2020 τι θα κάνουμε με τα άτομα αυτά. Γιατί ξέρουμε από την εμπειρία μας ότι όταν κάποιος έχει περάσει από μια τέτοια εκπαίδευση και από μια ρίζοσπαστικοποίηση και μένει στην επικράτειά μας, ε, θα είναι η βετεράνη του αύριο αυτή. Έχουμε και τα άτομα τα οποία έρχονται στην χώρα μας για να διαπράξουν τέτοιες επιθέσεις. Ε, τζιχαντιστές, ε, Ευρωπαίοι για παράδειγμα, που είναι κοντά στα σύνορα με την Τουρκία για παράδειγμα και κάποια μέλη εξ αυτών λοιπόν ε, απειλούν ε, τις, ε, την ασφαλειά μας εκπροσωπώντας το Ισλαμικό κράτος. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες αυτές. Τελευταίο σημείο σε ό,τι αφορά τις επιστροφές και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω το θέμα αυτό. Οι τζιχαλιστές αυτές οι Ευρωπαίοι αποτελούν αν θέλετε, συνάλλαγμα για πολλούς από αυτού του περιφερειακούς τομεί, ε, τι ένοπλε ομάδε ή τα κράτη, σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, ανταλλαγή με φυλακισμένου, σε ό,τι αφορά ε, τα σύνορα με τη Συρία, τα κράτη τα οποία με τη Συρία, όπου υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις ε, απέτηση για να επιστραφούν αυτά τα άτομα, να υπάρξουν συγκεκριμένε δράσει από τα ευρωπαϊκά κράτη. Τρίτο θέμα στο οποίο και θα κλείσω είναι η λειτουργική χρήση των ε, κοινωνικών ε, δικτύων στη φάση της ε, οργάνωσης και της εκτέλεσης δημοκρατικών επιθέσεων. Η συζήτηση για την προπαγάνδα που υπάρχει πραγματικά στο διαδίκτυο και έχει μεγάλη σημασία δεν θα πρέπει να σταματήσει γιατί έχουμε το θέμα αυτό της λειτουργικής χρήσης από, τέτοιες, από τέτοια δίκτυα που χρησιμοποιούν όλα αυτές τις υπηρεσίες του διαδικτύου για την προετοιμασία των χτυπημάτων. Και έγινε λοιπόν μια σχετική μελέτη από την ΚΑΤ για να εντοπιστούν οι διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να αποτρέψουμε την προπαρασκευτική αυτή χρήση του διαδικτύου. Και έχουμε διάφορα τέτοια παραδείγματα. Για παράδειγμα, στην επίθεση της 7ης Νοεμβρίου είχαν ε, Όλα αυτά προετοιμαστεί, είχε το χτύπημα στο Telegram χωρίς καμία χρήση ε, τηλεφώνου. Και η επίθεση στην Νέα Υόρκη ε, και στην New το 2016, όπου ε, η όλη η επικοινωνία των τρομοκρατών έχει γίνει μέσω Facebook. Νομίζω ότι στο μέλλον θα πρέπει να επικεντρωθούμε λοιπόν σε αυτού του τρει παράγοντε, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, από την πολιτική βούληση, η οποία σε πολλέ περιπτώσει ε, απουσιάζει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά το θέμα τη τρομοκρατία. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βρυζάρ, λέει πρόεδρο, για την ε, εντυπωσιακή αυτή παρουσίαση πραγματικά για το πώ έχει η κατάσταση σήμερα σε ό,τι αφορά την απειλή και τον ε, πολλαπλό χαρακτήρα τη απειλή ναι, ναι, ναι, 20 λεπτά, done. Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους με το λόγο που τον ζήτησε ο κ. Τανζόν για να ξεκινήσει. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ακούστε. Πιστεύω ότι η άσκηση επιτεύχθη. Είναι ενδιαφέρον να ακούμε το, το Brizard, γιατί μας ε, καλεί να σκεφτούμε τι θα κάνουμε. Βλέπουμε τις διάφορες ε, οπτικές γωνίες από όπου εξετάζουμε το θέμα, ενδεχομένως ιδέες που μπορεί να έχουμε. Αυτό που είναι σημαντικό βέβαια είναι η διάρκεια, κάτι το οποίο τόνισε και ο, και ο η διάρκεια ζωής των ε, οργανώσεων αυτών. Μπορούμε επίσης να δούμε τα πράγματα πιο ρεαλιστικά, χωρίς κάποιες υπερβολές που, που κάποιες φορές επηρεάζουν τη συζήτησή μας. Βλέπουμε ότι κάποια άτομα, όπως για παράδειγμα με την επίθεση που έλαβε χώρα πρόσφατα στη Γαλλία, κάποια άτομα δεν τα είχαμε υπόψη μας, δεν τους παρακολουθούσε κανείς. Πιστεύω ότι είναι ε, θεμελιώδες να ξέρουμε ότι κάποια άτομα δεν τα γνωρίζουν οι υπηρεσίες πληροφοριών. Και αυτό δεν είναι απλώς ένα πρόβλημα συντονισμού. Είναι επίση σημαντικό κάτι άλλο που δεν το ανέφερε σήμερα ο Μπρισσάρ, η, η χρηματοδότηση των τρομοκρατικών δικτύων. Είναι ανάγκη να έχουμε απτές αποδείξεις στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και στην χρηματοδότηση. Το Ισλαμικό κράτος έχει ένα ενδογενές πλέον σύστημα παρόμοιο με το σύστημα οποιοδήποτε κράτος που το επιτρέπει να αυτοχρηματοδοτείται. Αυτό που πρέπει να κάνουμε λοιπόν τώρα είναι να καταπολεμήσουμε την χρηματοδότηση αυτή. Πιστεύω ένα μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης των τρομοκρατικών αυτών οργανώσεων γίνεται μέσω οδών που μπορούμε να εντοπίσουμε. Το τελευταίο σημείο που θέλω να θίξω, κάτι το οποίο είναι πολύ σωστό, πέρα από τα νούμερα και τις στατιστικές, είναι το γεγονός ότι δεν μπορούμε να περιθωριοποιήσουμε την, την ιδεολογία. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε κυρώσεις στην ιδεολογία. Πίσω από όλες τις πράξεις υπάρχει μια ιδεολογία. Και αυτή την ιδεολογία δεν μπορούμε να τη μετρήσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, είναι κάπως ευρία η, η ερώτησή μου. Αλλά αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αν αυτή η ιδεολογία παραμένει τόσο δυνατή, τόσο, τόσο ισχυρή. αν αυτή η ιδεολογία μετατρέπεται σε πράξη μέσω της προπαγάνδας. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Αγνό Τάνσον. Δίνουμε άμεσα το λόγο στον Ζων Ζακ Πρίζα. Σε ό,τι αφορά τώρα την, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι ένα σύνολο πράξεων. Τα νούμερα υπάρχουν. Είναι δυστυχώς αρκετοί αυτοί που περνάνε από τη θεωρία στην πράξη, οι τρομοκράτε και δεν τους γνωρίζουν οι υπηρεσίες πληροφοριών. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειές μας, είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλοι εμείς, όχι μόνο οι, οι υπηρεσίες πληροφοριών. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση τώρα, αυτό το, το άρθρο των New York Times λέει ακριβώς αυτό ότι το Ισλαμικό κράτος ελέγχει μια ολόκληρη περιοχή. Σε αντίθεση με άλλες τρομοκρατικές εργανώσεις. Και αντλεί λοιπόν τους οικονομικούς του πόρους από αυτήν την γεωγραφική περιοχή την οποία ελέγχει. Και βεβαίως από την εκμετάλλευση των όλων των οικονομικών παραγόντων, των υπηκών, των πολιτών που ζουν στην περιοχή αυτή. Ενώ η Αλκάιδα, η το μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών πόρων που εισέρχονταν σε αυτήν την τρομοκρατική οργάνωση ερχόταν από εξωτερικούς παράγοντες, από εξωτερική χρηματοδότηση. Τώρα όμως μιλάμε για, ένα, για μια τρομοκρατική οργάνωση η οποία είναι αυτοχρηματοδοτούμενη κατά κάποιο τρόπο. Και αυτό είναι ο λόγος που δεν έχουμε λύση, δεν έχουμε τρόπο να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά τη χρηματοδότηση της ε, τρομοκρατικής αυτής οργάνωσης. προσπαθούμε, τα Ηνωμένα Έθνη πάγωσαν ένα μεγάλο μέρος ε, χρημάτων που κατευθυνόταν ε, προς το Ισλαμικό κράτος, αλλά δεν έχουμε βρει μια απόλυτη λύση για, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το, το νέο μοντέλο χρηματοδότησης. Πρέπει να βρούμε ένα τρόπο κυρώσεων κατά κάποιο τρόπο, χωρίς βεβαίως ε, να βλάψουμε τον ίδιο το το πληθυσμό των περιοχών αυτών. Η μάχη μας ενάντια στην τρομοκρατία είναι πολύπλοκη, πρέπει να μπορούμε να εντοπίζουμε την προέλευση των τζιχατιστών, για παράδειγμα. Κάτι το οποίο μπορούμε να το κάνουμε μέσω του ελέγχου της χρηματοδότησης. Να, να μπορούμε να εντοπίζουμε ε, τα διάφορα μοντέλα συμπεριφοράς. Ούτως ώστε να μπορούμε νωρίς να δούμε που προετοιμάζεται μια τρομοκρατική πράξη, για παράδειγμα, μια τρομοκρατική επίθεση. Πιστεύω ότι όλα μπορούν να είναι χρήσιμα, όλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ούτω ώστε να αποτρέψουμε τρομοκρατικές επιθέσεις. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ιδεολογίας τώρα, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι στα πλαίσια της τζιχαντιστικής λογικής αυτό που βλέπουμε είναι το γεγονός ότι χάνουν έδαφος τα παιδιά των μαχών κατά κάποιο τρόπο ενδυναμώνει την, την νομιμότητα τρόπων την ά των επιθέσεων εκτός των πεδίων μαχών. από πλευράς υποστηρικτών και μαχητών των τρομοκρατικών αυτών οργανώσεων, όπου προσπαθούν να, να στηρίξουν το, το μοντέλο αυτό των τσιχαντιστικών οργανώσεων. Βλέπουμε όλο και περισσότερο άτομα που φεύγουν από τη Συρία και το Ιράκ και μετατοπίζονται σε άλλες περιοχές, όπως σας είπα και πριν, στο Αφγανιστάν, στη Λιβύη και αλλού ούτως ώστε να εξακολουθήσουν να, να μάχονται υπέρ ε, της δρομοκρατικής οργάνωσης. Σας ευχαριστώ. Πολύ σαφής οι απαντήσεις ε, στην πληθώρα αυτή των ερωτήσεων. Η κυρία Γκόμες που είναι η συντονίστρια των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στην ομάδα. Σας ευχαριστώ. Κύριε ε, Μπριζάρ, μιλήσατε για τα 50 με 60.000 ριζοσπαστικοποιημένους και τον κατακαιρματισμό και την παγκοσμιοποίηση της τρομοκρατικής απειλής. Πέραν των προσπαθειών που μας περιγράψατε, προκειμένου να κινητοποιήσουμε και τους τοπικούς φορείς, ε, πώς μπορούμε να κινητοποιήσουμε τους δικούς μας μουσουλμάνους, τους μουσουλμάνους ε, των δικών μας χωρών, γιατί χωρίς τη δική τους εμπλοκή είμαστε χαμένοι από χέρι δεν θα πρέπει να του αφήσουμε βορρά στον ελιτισμό των Βουαχαμπιτών ε, ή στον αντισλαμισμό, στην ισλαμοφοβική συμπεριφορά κάποιων λαϊκιστικών δυνάμεων ή κάποιων ε, κοινωνικών στρωμάτων ε, ή στο έρμεο των δημαγωγών. Επίσης, έχουμε εκατοντάδες φυλακισμένους Ευρωπαίους ε, θα τους αφήσουμε στην κουρδική ζώνη. Θα τους αφήσουμε να γίνουν θύματα των ε, Τούρκων. Γιατί ε, δεν αφήνουμε καν τους Κούρδους να αντιμετωπίσουν αυτούς τους Ευρωπαίους φυλακισμένους που πήγαν εκεί τελικά τι για να κατασφαγιαστούν. Επίσης, τι γίνεται με την απειλή που προέρχεται από τη Λιβύη με, το, με τη σύγχυση που δημιουργήθηκε εκεί. Επίσης, ε, ε, θα μιλήσουμε και αυτό αργότερα με τον κύριο Μοσκοβισή, αλλά μιλήσαμε για 10 δισεκατομμύρια από, τις, ε, από τους ειδικούς φόρους του κατανάλωση και 50 δισεκατομμύρια από την απάτη με το ΦΠΑ που ξέρουμε ότι και εδώ και καιρό γνωρίζουμε ότι χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας αυτά τα κονδύλια ή για τη χρηματοδότηση εγκληματικών κυκλωμάτων που έχουν σαφείς διασυνδέσεις με τρομοκρατικές οργανώσεις και με την Αλκαϊδα. Ενώ οι κυβερνήσεις φαίνεται ότι διαφορούν και δεν μπαίνουν καν στον κόπο να θεσπίσουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Τι γνώμη έχετε για τον τρόπο ε, χρηματοδότηση των τρομοκρατικών οργανώσεων από το δικό μας το σύστημα, από τα, τις δικές μας αδυναμίες και από την απροθυμία των κυβερνήσεων να ρυθμίσουν αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Πολλέ είναι οι ερωτήσει και τεχνικέ αλλά και πολλέ πολιτικέ ε, ερωτήσει έγιναν από την κυρία Γκόμε. Ναι, ευχαριστώ. Γνωρίζω θαυμάσια τον τρόπο μικροχρηματοδότηση των τρομοκρατικών οργανώσεων, γιατί μιλήσαμε πριν για τη μακροχρηματοδότηση, αλλά έχουμε και τη μικροχρηματοδότηση. Αυτό που παρατηρούμε και για το θέμα αυτό, ε, γιατί μίλησα για τη μακροχρηματοδότηση πριν και για το γεγονός ότι σήμερα το μοντέλο των κυρώσεων ε, ήταν αναποτελεσματικό, ήταν ακατάλληλο για τον τρόπο, το μοντέλο της μακροχρηματοδότησης, αλλά έχουμε και τη μικροχρηματοδότηση. Και τα μέτρα μας προσπαθούν να μειώσουν τον αντίκτυπο κάποιων ε, μέσων που χρησιμοποιούν οι τρομοκράτες. Για παράδειγμα, επικεντρωθήκαμε στην κρυπτογράφηση. Είπαμε ότι χρησιμοποιούν κρυπτογραφημένα μέσα, ε, κρύβονται, κρατούν την ανωνυμία τους. Αλλά όχι μόνο. Είδαμε ότι οι τρομοκράτες και από τις επιθέσεις των ε, Βρυξελών και του Παρισιού ότι χρησιμοποιούν και νόμιμους διάβλους επικοινωνία και πληροφόρηση, αλλά με ανώνυμο τρόπο. Και αυτή η δυνατότητα να κρατούν την ανωνυμία του ό,τι αφορά τη μεταφορά κονδυλίων, τα εμβάσματα, ε, δεν έχει επιληθεί για πολλούς και διάφορους λόγους. Πάντως οι, οι τρομοκράτες χρησιμοποιούν αυτά τα κενά του συστήματός μας για να χρηματοδοτηθούν. Το είδαμε και με τις ε, προπληρωμένες ε, πιστοτικές κάρτες, μάλλον τις προπληρωμένες κάρτες. Χρησιμοποιούνται μαζικά αυτές οι προπληρωμένες κάρτες από όλη την αλυσίδα ό,τι υπόθεση τρομοκρατική να πάρουμε, διαπιστώνουμε συστηματική χρήση των προπληρωμένων καρτών. Και τι κάνουμε, τίποτα. Μειώνουμε απλώ το ανώτοτο όριο για τη χρήση του, για τι πληρωμέ. Αλλά δεν επιλύουμε το, το πρόβλημα στη ρίζα του. Και το πρόβλημα είναι η δυνατότητα της ανωνυμίας, γιατί οποιοδήποτε μπορεί να αγοράσει από ένα περίπτερο ε, μια προπληρωμένη κάρτα και να τη χρησιμοποιήσει για να αγοράσει υλικό συστατικό για να δημιουργήσει ένα αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό ή να μετακινηθεί, να χρησιμοποιήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή να νοικιάσει ένα διαμέρισμα για να αναπτύξει τι δραστηριότητέ του και ούτω καθεξής. Η ανωνυμία είναι το πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν να προσαρμόσουμε την καταστολή μα στη νέα πραγματικότητα, αλλά δυστυχώ εμεί στερούμε. Εμεί τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε, γιατί είναι πολύ πιο γρήγοροι οι τρομοκράτε και αξιοποιούν αυτά τα κενά. Σε ό,τι αφορά τη Λιβύη. Για τη Λιβύη το είπα ότι διαπιστώνουμε πως ε, οι Ευρωπαίοι πηγαίνουν, ε, μέσω της, πηγαίνουν στη Λιβύη και εκεί προσχωρούν στο Ισλαμικό κράτος. Και σήμερα το χάος είναι λιγότερο από ό,τι πριν από μερικά χρόνια. Αλλά αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι ε, σταδιακά η κατάσταση στη Λιβύη και κυρίως στην Τινησία ε, εξαπλώνεται στην ευρύτερη περιοχή. Και κάποιες κυβερνήσεις της υποσαχαρίου Αφρικής ε, ανησυχούν από την επιστροφή τζιχαντιστών στις χώρες αυτές. Οπότε υπάρχει μια μεγάλη βεβαιότητα για το μέλλον. Και τα μέσα που έχουμε εκεί δεν είναι τελείως ακατάλληλα για την ε, τοπική πραγματικότητα. Και και οι μυστικές υπηρεσίε και τα στρατιωτικά μέσα είναι ελάχιστα και πενιχρά. Γι' αυτό η Γαλλία και άλλες χώρες έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν εκεί μακροπρόθεσμα στις χώρες αυτές δηλαδή για να εξασφαλίσουν και τη δική του ασφάλεια και να εγγυηθούν ε, την, την ασφάλεια γιατί είχαμε λαθρεμπόριο όπλων, βαρέων όπλων από τη Λιβύη προ άλλε χώρες. Θα πρέπει να παρεμποδίσουμε και να εξαλείψουμε τέτοιου είδους παράνομων κινήσεων λαθρεμπόριο όπλων. Σε ό,τι αφορά τις επιστροφές τι είπατε. Τους Ευρωπαίους κρατουμένους. Ναι, κάποιοι Ευρωπαίοι τζιχαντιστές είναι φυλακισμένοι σε, και κρατούνται από τους Κούρδους της Συρίας που είναι ένοπλη δύναμη και δεν υπάρχει καμία υποχρέωση ε, δίκης ε, της ε, χώρας προέλευσης των ε, ανθρώπων αυτών. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, ε, εδώ η τοπική δικαιοδοσία υπερισχύει. Η δοσηδικία δηλαδή. Οπότε δεν θα πρέπει να μπούμε σε μια λογική διαπραγμάτευσης με τις κουρδικές ενόπλες δυνάμεις, γιατί αυτοί οι τσιχαντιστές ε, σήμερα είναι το αντικείμενο σημαντικό παζαρεμάτων που γίνεται Και κατά τη γνώμη μου θα ήταν επικίνδυνο να εμπλακούμε σε αυτό το παζάρεμα. Και τώρα, τι γίνεται με τη, την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου στην επικράτεια εκείνη. Μα δεν ασχολούνται με αυτό οι Κούρδοι. Οι Κούρδοι ασχολούνται τώρα με τον πόλεμο. Και υπάρχουν και κάποια, ε, κάποιες άλλες ομάδες ε, ενοπλές στη Συρία που ίσως θα διεκδικήσουν την αρμοδιότητα για την ε, δίκη αυτή, εφόσον φυσικά το δικαστικό σύστημα εξασφαλίζει τα απαραίτητα δικονομικά εχέγγυα τη δίκαιη δίκη και ούτω καθεξή. Επίσης έχουμε ένα άλλο φαινόμενο, δεν ακούσαμε εκτό μικροφώνου το σχόλιο της κυρίας Γκόμενες, της κυρίας ε, για την εμπλοκή των μουσουλμανικών κοινότητων στις χώρες μας. Όντω πολλέ κοινότητε. Ε, ε, έχουν, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο αυτό κάπως τους ξεπερνά και είπατε να εμπλέξουμε τις τοπικές κοινότητες αλλά να εμπλέξουμε και ε, τις μουσουλμανικές κοινότητες. Το θέμα είναι τι περιμένουμε από αυτές τις μουσουλμανικές κοινότητες γιατί μερικές φορές ε, όταν μιλούμε συγχαίουμε πολλά πράγματα και το αμάλγαμα μπορεί να είναι εύκολο ή να πούμε, ας πούμε ότι όλες, ε, όλοι οι σαλαφίστες είναι και τζιχαντιστές. Αυτό όμως είναι λάθος, γιατί είδαμε ότι και ανάμεσα στα αυτά τα δύο ρεύματα, τζιχαντιστών και σαλαφιστών, υπήρχαν τεράστιες διαφορές, στην Αλγερία και αλλού. Οπότε η υπεραπλούστευση δεν είναι καλή, τζιχατιστες αυτο είναι πολύ πιο περίπλοκα τα δυο ρευματα τζιχατιστων και σαλαφιστων υπηρχαν τεραστιες διαφορες στην αλγερια και αλλου οποτε η υπεραπλουστευση δεν ειναι καλη γιατι ειναι πολυ πιο περιπλοκα τα πραγματα και οι σαλαφιστές απορρίπτουν ε, τον τζιχαντισμό. Παρόλο που μπορεί να πηγάζουν και τα δύο ρεύματα από την ίδια βάση, έχουν διαφοροποιηθεί έντονα. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε σπευσμένες και βεβαιασμένες αναλύσεις για περίπλοκα φαινόμενα και κυρίως να μην κατηγορούμε αβάσιμα. Επίσης, έχουμε κάποιους που, για τους οποίους η τρομοκρατία είναι τρόπος δράσης ε, και μετατρέπουν την τρομοκρατία σε ιδεολογία και σε στρατηγικό του στόχο. Βέβαια, έχουν... αυτός είναι ένας τρόπος δράσης κυρίως τελικά η τρομοκρατία. Και δεν θα πρέπει να στιγματίζουμε ολόκληρες κοινότητες επειδή κάποια μέλη τους α, έχουν τρομοκρατική δράση. Σας ευχαριστώ, λέει και πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις απαντήσεις στα τέσσερα αυτά ερωτήματα. Ε, σημαντικά στα θέματα, τα οποία προφανώς και μένουν σε ένα βαθμό ανοιχτά ακόμα. Να δώσω το λόγο στον κύριο Ζεράτεπρε από την Άλντα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και καταρχάς, ε, να συμφωνήσω με τους συναδέλφους που εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για την παρουσίαση που ακούσαμε. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ σαφής και ξεκάθαρη. Εμένα αυτό που με απασχολεί ιδιαίτερα κύριε Μπριζάρ είναι να μάθουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως έχει. Γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ε, στοιχεία στα οποία θα πρέπει να ανταποκριθούμε, θα πρέπει να θέσουμε στόχους και στην Επιτροπή μας εδώ, σε αυτήν την Ειδική Επιτροπή. Έχω τρεις-τέσσερις ερωτήσεις λοιπόν να, να σας απευθύνω σε λειτουργικό επίπεδο. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της απειλής, η υπεύθυνη ασφαλεία σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα συναντιόνται σε, κάποιο, σε κάποια πλατφόρμα για να συζητήσουν τη διαμόρφωση της, ε, και την εξέλιξη των απειλών, το πόσο κατεπήγουσε είναι και ούτω καθεξής η Ευρωπόλου Η Ευρωπόλ παίζει ή θα μπορούσε να παίξει πιο σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό. Μιλάμε για ριζοσπαστικοποίηση. Μα είπατε αρκετά ανησυχητικά στοιχεία. 50 έως 60 χιλιάδες ριζοσπαστικοποιημένη στην ε, Ευρώπη. Το διπλάσιο του βαλγικού στρατού. Εντάξει, δεν είναι και πιο μεγάλο στρατό τη Ευρώπη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Όλα αυτά τα άτομα προφανώ δεν προβούν απαραίτητα σε επιθέσει, αλλά υπάρχουν ανταλλαγέ πληροφοριών μεταξύ των διάφορων μυστικών υπηρεσιών σε ό,τι αφορά τα στοιχεία τα οποία θα μας υποδείκνυαν ε, ενδεχόμενη επίθεση το κατά πόσον είναι πιθανόν ή όχι. Πώς θα μπορούσαμε δηλαδή να βάλουμε στο στόχο τα άτομα τα οποία είναι υψηλής επικίνδυνοτητας και να κάνουμε πιο καλές ε, μελέτες. Στη χώρα μου, στο Βέλγιο, δεν επικοινωνούμε και δεν λέμε στους δημάρχους ε, δεν, είμαστε είμαι ο δημάρχους σε ό,τι αφορά ενδεχόμενε τρομοκρατικέ απειλέ στην περιφερειά τους, για να μην υπάρχει κίνδυνο ε, πανικού. Τι προτείνεται λοιπόν να γίνει σε τοπικό επίπεδο σε ό,τι αφορά του κανόνες που ενδεχομένω υπάρχουν, τις πρακτικές που ακολουθούνται. Ύστερα, για τα μέσα κοινωνική δικτύωση, ακούσαμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσατε. σε ό,τι αφορά τα θέματα κρυπτογράφηση, ε, πώ αντιμετωπίσετε τα προβλήματα αυτά τα τελευταία χρόνια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τέλος, ε, μου κάνει εντύπωση που σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει καμία εναρμόνιση σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό επίπεδο τη απειλή. Ε, στη Γαλλία έχουμε επίπεδο 3, για παράδειγμα. Στην Γαλλία 4, αν δεν κάνω λάθο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ενδεχομένω να υπάρχει άλλο επίπεδο επικινδυνότητας σε ό,τι αφορά ενδεχόμενη απειλή υπάρχει κάποια εναρμόνιση και του επίπεδου του κινδύνου, αλλά και των μέτρων που ακολουθούνται σε κάθε επίπεδο. Μήπως, ε, γιατί σε κάθε χώρα υπάρχουν πρωτόκολλα και μήπως θα ήταν ευκταίο να υπάρχει μια συντονιστική δράση στα επίπεδα αυτά και στις, στα μέτρα αυτά. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, πολύ ενδιαφέροντα τα ερωτήματα που μα θέσατε. Το θέμα τη αξιολόγηση ε, τη άπειλης. Ε, γιατί γιατί αυτό είναι το βασικό σας ερώτημα που δεν καταλαβαίνω. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε εκπρόσωποι εδώ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προφανώς. Το πρόβλημα είναι το εξή. Συχνά αναρωτιέμαι γιατί δεν προχωράμε πιο γρήγορα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη κινητοποίηση από το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και των άλλων από τα άλλα θεσμικά όργανα. Γιατί αν σκεφτούμε ότι μας χρειάστηκαν 12 χρόνια για να καταλήξουμε για ένα, σε ένα κείμενο για το PNR σε ό,τι αφορά μεγάλες τρομοκρατικές επιδύσεις στην ε, ε, Μαδρίτη το 2004-2016 στις Βρυξέλλες. Χρειάστηκαν λοιπόν δύο τέτοια, δύο, τέτοια μεγάλα τρομοκρατικά χτυπήματα για να καταλήξουμε επιτέλους σε ένα κείμενο για το PNR. Το οποίο αποτελεί και μία μόνο συνιστός, αν θέλετε, του προβλήματος. Ένα μόνο στοιχείο στο σύνολο του φαινομένου αυτό είναι ο πυρήνα του προβλήματο ουσιαστικά, γιατί τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν την ίδια αντίληψη ε, τη ε, τρομοκρατική απειλή. Μου έκανε εντύπωση, γιατί συμμετείχα σε ένα συνέδριο πρόσφατα με έναν πρώην Υπουργό Εξωτερικών, με έναν, ε, από, με έναν Υπουργό Εξωτερικών, πρώην Υπουργό Εξωτερικών μια χώρα τη Ανατολική Ευρώπη. Και στην παρέμβαση του τι δήλωσε ουσιαστικά σε ένα συνέδριο για την τρομοκρατία, θεωρούμε ότι η χώρα μας δεν αποτελεί στόχο τρομοκρατών και άρα για μας δεν μας απασχολεί ιδιαίτερος και καταραπατριάζεται το θέμα αυτό. Πήρα το λόγο και απάντησα ότι κοιτάξτε, λάθος κάνατε, γιατί το γεγονός ότι η χώρα σας δεν έχει αποτελέσει ακόμα ε, στόχο δεν σημαίνει ότι δεν αποτελεί κέντρο και χώρα διαμετακόμισης και διέλευσης των τρομοκρατών. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι δεν έχουμε όλοι την ίδια αντίληψη για τον κίνδυνο και τις απειλές. Άρα, όταν καλούμαστε να πάρουμε κοινέ αποφάσεις, ε, χωλένει η κατάσταση. Σε ό,τι αφορά το θέμα της ανταλλαγής πληροφοριών, ναι, υπάρχουν ανταλλαγές καθημερινές. Σε ό,τι αφορά απειλέ, σε ό,τι αφορά ενδεχόμενα επικίνδυνα άτομα και προφανώς η Ευρωπόλη θα πρέπει να δραματίσει σημαντικό ρόλο. Ασφαλώς. Γιατί ακόμα και σήμερα, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, παρά τα μέτρα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, πιστώνουμε ότι θα πρέπει να είναι πολύ πιο λειτουργικό το σύστημα από ό,τι είναι στην παρούσα φάση. Και η Ευρωπόλ και η Eurojust αποτελούν ε, υπηρεσίε διευκόλυνση ε, και θα πρέπει προφανώ να παίξουν όλο και μεγαλύτερο ρόλο σε λειτουργικό επίπεδο. Θεωρώ ότι οι ερωτήσεις σας είναι πιο πολύ πολιτικής φύσεως. Αυτό είναι το θέμα, ότι αν θέλουμε να προχωρήσουμε από κοινού θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάποια βασικά πράγματα. Σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την, ε, το επίπεδο του κινδύνου, είτε αφορά το συντονισμό για την αντιμετώπιση των επουλών, είτε οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή αντίληψη για τον κίνδυνο και την απειλή σε πρώτη φάση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εμπλοκή του τοπικού επίπεδου, αυτό γίνεται σε κάποιες περιπτώσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις ε, τα προγράμματα στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γερμανία. Υπάρχουν τέτοια προγράμματα κινητοποίησης του τοπικού επίπεδου. Αλλά αυτό αφορά και ένα μόνο, ένα μόνο παράγοντα. Το θέμα το κοινωνικό, το θέμα το, της εκπαίδευσης, της παιδείας. Ε. Χρειαζόμαστε όμως και τη συμμετοχή των ε, τοπικών ενώσεων, των κοινωνικών ενώσεων, των θρησκευτικών ενδεχομένω ε, φορέων, για να υπάρχει συζήτηση μεταξύ των φορέων αυτών, να υπάρχει συνεργασία μεταξύ όλων αυτών των φορέων για καλύτερη ενημέρωση, να υπάρχει καλύτερος διάλογος, να εντοπίζονται τα συμπτώματα, να εντοπίζονται οι αδύναμοι κρίκοι και να αναλαμβάνει κάθε φορέα στην ευθύνη του, γιατί προφανώς σήμερα Μπορεί να υπάρχει κάποια εκπαίδευση, κάποια κατάρτιση, αλλά τίποτα συστηματικό. Θα πρέπει να υπάρχει πολύ πιο συστηματική αντιμετώπιση και δεν σας μιλώ μόνο για την ενημέρωση, σας μιλώ και για την ε, πρόληψη, την ε, λειτουργία, την, ε, το σχηματισμό τέτοιων πυρήνων για να εντοπίζονται τα άτομα τα οποία αποτελούν κίνδυνο. Να δούμε και ποιες θα είναι οι απαντήσεις, ποια θα είναι η αντίδραση που θα πρέπει να δίδεται σε ό,τι αφορά τέτοια επικίνδυνα άτομα τα οποία αποτελούν κίνδυνο. Να υπάρξει μια πραγματική κινητοποίηση, το οποίο δεν ισχύει δυστυχώ σήμερα. Για τα εργαλεία και τα εργαλεία της κοινωνικής δικτύωσης, ε, ναι. Το θέμα τη κρυπτογράφηση. Αυτό έχει απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε προχωρήσει με πολύ κόπο. Υπάρχει και ευρωπαϊκός ε, συντονιστής σήμερα. Το θέμα, για παράδειγμα, ότι έχουμε περάσει σε επίπεδο ε, που υπάρχει η λειτουργική χρήση των εργαλείων αυτών και από τους ε, τρομοκρατών, νομίζω ότι έχει μεγαλύτερο αντικτύπο από ότι, για παράδειγμα, η προπαγάνδα, γιατί ξέρουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις προστατεύονται οι υπεύθυνοι προπαγάνδα από το εθνικό δίκαιο. Εδώ μιλάμε για συμμετοχή, πραγματική συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα, τα οποία επιτρέπουν τελικά σε κάποιες φορείς να διαπράττουν τρομοκρατικά χτυπήματα. Και όπω σα είπα, σε πολλέ περιπτώσει, χωρί τα εργαλεία αυτά δεν πρόκειται να είχαν πετύχει οι τρομακτικέ αυτέ επιθέσει. Δεν υπήρχε περίπτωση. Και έτσι βλέπουμε πόσο σημαντικά είναι. Και αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να. Ε, το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι ότι θα πρέπει να αναλάβουν όλη την ευθύνη του και στο διαδίκτυο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπριζάρ. Ο κύριο ε, Ντεπρέ μίλησε για 60.000 άτομα τα οποία είναι παστικοποιημένα. Είπα μεταξύ 50 και 60 ε, χιλιάδων, ναι, διπλάσια από τον ε, βελγικό στρατό. Προτού τόσο το λόγο στον κύριο Φανόρντεν, ε, θα μπορούσα να σας ζητήσω να μας κάνετε μια συντομή ανάλυση των στοιχείων αυτών, αστρονομικών πραγματικά. Ο κύριος Ντανζόν μας μίλησε για την ε, επίθεση την οποία πετράπηκε στη Γαλλία. Μιλήσατε για τα ριζοσπαστικοποιημένα άτομα τα οποία θα βγουν από τη φυλακή, θα εκτίσουν την ποινή του, θα ολοκληρώσουν την έκθεση τη ποινή του, θα του παρακολουθήσει αυτού η αστυνομία. Τι θα γίνει και τι γίνεται και με αυτά τα 50-60 χιλιάδε άτομα τα οποία έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί. Να δώσω το λόγο στον κύριο Βαν Όρντεν και θα μου απαντήσετε αν θέλετε και εμένα στη συνέχεια. Και τρίτη σύντομη ερώτηση, μια και έχω το μικρόφωνο. Ακούσαμε ότι ο Μπασάμα Γιασί πρώην τρομοκράτης πάνω από 60 χρονών, 71 χρονών, ε, πέρασε από την Ευρώπη χωρίς κανένα πρόβλημα πρόσφατα τον συλλάβανε κάπου κοντά στην ε, Τουρκία. Ενδεχομένω να έχει βγει στη σύνταξη, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάπω προκλητικό αυτό ω γεγονό. Να δώσω το λόγο στον κύριο Φανόρντεν από το Ηνωμένο Βασίλειο. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τον κύριο Πρίζα για, τις... για την παρουσίασή του. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της κοινή απειλή, δεν πιστεύω ότι αυτό είναι ένα θέμα εθνικών κυβερνήσεων. Υπάρχουν πάμπολοι μηχανισμοί που μπορούν να μας βοηθήσουν να έχουμε μια κοινή αξιολόγηση. Υπάρχει η Europol, υπάρχουν αντιτρομοκρατικές επιτροπές. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της απειλής. Το πρόβλημα για μένα σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση είναι η διαφορά μεταξύ αριστερά και δεξιά για να κάνουμε έτσι, να δώσουμε και μια πολιτική διάσταση. Αυτό έχει να κάνει και με το PNR. Για παράδειγμα, δεν είχε να κάνει με τις εθνικές κυβερνήσεις. Ουσιαστικά ήταν ε, ένα θέμα διαφορετικής αντίληψης από διαφορετικές πολιτικές ομάδες. Και ήθελα απλώς να κάνω αυτό το σχόλιο. Έχω καμία-δύο ερωτήσει. Μιλήσατε διεξοδικά για τους ε, τζιχαντιστές που επιστρέφουν και είμαστε λίγο μπερδεμένοι. Δεν ξέρουμε πώς ακριβώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό. Μας είπαν ότι κάποιοι συλλαμβάνονται και διώκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε αυτό το πρόβλημα με άτομα που είναι ύποπτα για δολοφονίες και δεν είμαστε... Δεν ξέρουμε τι ακριβώ πρέπει να κάνουμε με αυτές τις ομάδες ατόμων που έχουν μια πράξη εγκλήματα. Αναρωτιέμαι μήπως υπάρχει κάποια, κάποιο διεθνές δικαστήριο που θα έπρεπε να αντιμετωπίζει τα προβλήματα αυτά, τα άτομα αυτά. Ε, μετά υπάρχει το ζήτημα της ποινή, αν θα πρέπει να υπάρχουν ειδικέ εγκαταστάσεις για αυτά τα άτομα. Έχουμε και εμείς παραδείγματα. Είναι προβληματικό το σημείο αυτό. Υπάρχει μια θεμελιώδης ερώτηση, ένα θεμελιώδης ζήτημα το οποίο πρέπει να σκεφτούμε. Η έτερη ερώτησή μου έχει να κάνει με το κατά πόσο θα πρέπει να μας ανησυχούν τα όπλα μαζικής καταστροφής σε σχέση με την τρομοκρατία. Θα πρέπει να μας απασχολεί μια κυβέρνηση στην οποία μπορεί να έχουν εισχωρήσει τρομοκρατικά στοιχεία κατά κάποιο τρόπο. Βεβαίως ανησυχούμε για αυτοκίνητα που πραγματικά πατάνε τον κόσμο, τρέχουν και πατάνε πεζούς και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Αλλά αν ξεκινήσουμε την κουβέντα για όπλα μαζικής καταστροφής, ε, τότε περνάμε σε τελείως διαφορετικό επίπεδο. Δεν ξέρω ποιες είναι οι σκέψεις σας πάνω σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Μπριζάχ. Πρώτα απ' όλα να απαντήσω στην πρόεδρο σε ό,τι αφορά αυτά τα 50 με 60.000 άτομα. Αυτά είναι στατιστικά στοιχεία που προέρχονται από διάφορες κυβερνήσεις. Είναι εκτιμήσεις που έχουμε για άτομα που έχουν ρίζος παστικοποιηθεί. Κάθε χώρα βεβαίως έχει τη δική της, το δικό της ορισμό σχετικά με το τι είναι ένα ρίζος παστικοποιημένο άτομο. Αυτά όμως είναι τα συγκεντρωτικά στοιχεία που έχουμε από όλε τις χώρες σε ό,τι αφορά, επαναλαμβάνω, τα ριζοσπαστικοποιημένα άτομα. Τώρα σε ό,τι αφορά τα επικίνδυνα άτομα που ακολουθούνται από τις υπηρεσίες, έχουμε να κάνουμε με 10.000 άτομα. Αυτά είναι άτομα που είναι ε, δυνητικά επικίνδυνα. Σε ό,τι αφορά τώρα το ερώτημα της παρακολούθησης από πλευράς υπηρεσιών πληροφοριών, ε, έχουμε πολλαπλές στρατηγικές, τακτικές που ακολουθούμε έχει να κάνει με την προσοχή μας η οποία θα πρέπει να είναι στραμμένη σε αυτά τα άτομα. Η παρακολούθηση είναι παρακολούθηση από απόσταση θα έλεγα διακριτική έντοση εισαγωγικών ε, παρακολούθηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ε, συλλογή των ε, μηνυμάτων που ανταλλάζουν των ηλεκτρονικών δεδομένων και στη συνέχεια ανάλυση όλων των στοιχείων αυτών. Δεν έχω στοιχεία συγκεκριμένα σχετικά με το πόσα τέτοιου τύπου δυνητικά άτομα παρακολουθούνται, αλλά η παρακολούθηση μπορώ να σας πω ότι έχει διαφορετικά εργαλεία, διαφορετικές τεχνικές. Σε ό,τι αφορά τώρα τα μεμονωμένα, τις μεμονωμένες περιπτώσεις ατόμων που βρίσκονται στις ε, Βρυξέλλες ή και στην Γαλλία. σε ό,τι αφορά τους θρησκευτικού πυρήνες σε διάφορες περιοχές. Βεβαίως, ε, εκεί πέρα θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή από πλευρά των αρχών. Υπάρχει ένα σχολείο μικροφώνου. μικροφόνου. Εσείς τώρα, κύριε, με ρωτήσατε για το PNR. Υπάρχουν χώρες που αντιτίθεται σε αυτό το, το ζήτημα α, αξιοποίησης προσωπικών δεδομένων. Είναι ένα, είναι ένα ζήτημα πολιτικό, είναι ένα ζήτημα εθνικής θέσης σε πολλές περιπτώσεις. Κάποιες χώρες γιατί δεν έχουν αποτελέσει στόχο των τρομοκρατών, δεν έχουν απαραίτητα την ίδια οπτική γωνία που έχουμε εμείς. Υπάρχουν χώρες που δεν συντάσσονται με την λογική ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων. Σε ό,τι αφορά τώρα το διεθνέ Δικαστήριο, ναι, θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική ιδέα να υπάρχουν αρμόδια διεθνή δικαστήρια όπου θα πρέπει και θα μπορούν να δικάζονται αποτελεσματικά οι τζιχαντιστές και να καταδικάζονται για τα εγκλήματα πολέμου που έχουν διαπράξει. Είναι μια εξαιρετική ιδέα. Και να μην είναι στην αρμοδιότητα των εθνικών, των τοπικών δικαστηρίων τα εγκλήματα αυτά, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχει όμως μια πολιτική συνοχή, δεν υπάρχει μια πολιτική σύνεση σε αυτό το, το ζήτημα. Υπάρχουν ενστάσεις από διάφορα κράτη. ό,τι αφορά τώρα τα όπλα μαζικής καταστροφής και την τρομοκρατία. Αυτό είναι ένα αστικό μύθος, ε, θα λέγαμε, αποτελεί μέρος ενός αστικού μύθου. Έχουμε κάποιες ποραδικές πληροφορίε. δεν έχουμε όμως δει ποτέ σε επιχειρησιακό επίπεδο τρομοκρατικές οργανώσεις να ακολουθούν τέτοιες ε, τακτικές. Πάντοτε δίνω ένα παράδειγμα που για μένα είναι ιδιαίτερα ενδεικτικό αφορά στην 11η Σεπτεμβρίου. Το αρχικό σχέδιο δεν ήταν να χτυπήσουν τους, τους δίδυμους πύργους. Αρχικά θέλανε να ρίξουν τα αεροπλάνα σε ε, πυρηνικούς αντιδραστήρες. και ο Μπιν Λάντεν ε, πρώτος είχε την, την ιδέα. Ε, βεβαίως τέθηκε πιτάπιτο το ζήτημα των παραγόντων που δεν μπορούσαν να υπολογίσουν. Στόχος τους βεβαίως ήταν να πλήξουν ως το δυνατόν μεγαλύτερη μερίδα πληθυσμού Επομένω, η ιδέα που έπεσε στο τραπέζι ήταν ακριβώς αυτό που συνέβη, να ρίξουν τα αεροπλάνα στου ε, δίδυμου πύργου. Και το σχέδιο το, το αποδέχτηκαν. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι βεβαίως οι τρομοκρατικές οργανώσεις έχουν πειραματιστεί με διάφορους τρόπους αρκετοί τρομοκράτες έχουν τραυματιστεί και ήδη και ίδιοι χωρίς να φέρουν μεγάλα πλήγματα στον γενικό πληθυσμό. Προφανώς αυτού του τύπου οι επιθέσεις είναι μάλλον ιδιαίτερα πολύπλοκες για αυτού του τύπου τις τρομοκρατικές οργανώσεις οι τρομοκρατικέ οργανώσεις είναι μάλλον καιροσκοπικέ οργανώσεις. Έχουν ένα πολύπλοκο σύστημα δράση, το βλέπουμε καθημερινά, αλλά στόχος του είναι να δρουν όσο δυνατόν πιο αποτελεσματικά, γρήγορα και άμεσα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν εγώ δεν θεωρώ ότι οι τρομοκρατικές οργανώσεις θα μπορούσαν να κάνουν, να φέρουν τέτοιου τύπου χτυπήματα με όπλα μαζικής καταστροφής. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στις δύο συνεισηγήτριές μας, την κυρία Μόνικα Χολμάγερ και την κυρία Χέλγα Στίβενς. Μετά θα ακούσουμε δύο ακόμη συναδέλφους και θα ολοκληρώσουμε αυτό το σκέλος της συζήτησης. Κανονικά μέχρι τις 4.30. Όλγα και Κριστίν Βιλμέρκ μετά τις δύο συνεισηγητές. Πρώτα όμως η Μόνικα Χολμάγερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και τον κύριο Μπριζάρ για το γεγονό ότι έχουμε την ευκαιρία σήμερα να συζητήσουμε μαζί σας. Στα εισαγωγικά έχω μείνει, μέχρι να βάλετε τα ακουστικά σας. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι για τη σημερινή μας συζήτηση. Και για να ξεκινήσω από το τελευταίο σημείο για μένα ως εισηγήτρια και συνεισηγήτρια, τα σχόλια είναι πολύ διαφορετικά. Η Βρετανική κυβέρνηση, για παράδειγμα, εκφράζεται διαφορετικά σε σχέση με την, Αγγλική, σε σχέση με την Γερμανική και Γαλλική ε, κυβέρνηση. Αυτό προφανώς δεν απλοποιεί τα πράγματα, αλλά να πω το εξή. Ο κοινό παρανομαστής είναι σε ό,τι αφορά τα όπλα μαζική καταστροφή ε, είναι σαφή η δήλωση και οι δηλώσει ε, θα πρέπει να υπάρξει δηλαδή προληπτική ε, δράση προκειμένου να μην έχουν πρόσβαση σε υλικά τα οποία δεν πρέπει να έχουν στα χέρια τους. Είτε πρόκειται για πυρηνικά, είτε πρόκειται για βιολογικά, για χημικά. τα συστήματα ανιχνευσιμότητα, τα συστήματα πρόληψης, τα συστήματα όλα αυτά θα πρέπει να φροντίσουν προκειμένου να μην μεταφέρονται στα σύνορά μας ε, με ανεξέλεκτο τρόπο κάποια υλικά. Αυτό θεωρώ αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα. Γιατί δεν θα θέλαμε φυσικά να προκαλέσουμε ε, πανικό με το θέμα των όπλων μαζικής καταστροφής. Ένα δεύτερο ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει με, την, ε, με τις εθνικές κεντρικές ε, μονάδες, την κεντρική ή τοπική διαμόρφωση της μας. Το αναφέρατε, αναφέρετε το θέμα των ΜΚΟ, των δημάρχων, της τυπικής διάστασης. Να σας πω ότι γίνεται, έχει γίνει μία συζήτηση γιατί φαίνεται ότι κάποιοι είναι οι καλοί ή κάποιοι όπως η αστυνομία είναι οι κακοί, άσπρο μαύρο. Το θέμα είναι όμως και οι δύο πλευρές να έχουν πλήρης εμπιστοσύνη και να υπάρχει και αμοιβαία ενημέρωση και πληροφόρηση και οι κοινωνικές λοιπόν αρχές να ενημερώνουν την αστυνομία και αντίστροφα. Το ίδιο ισχύει και για τις ΜΚΟ, γιατί συχνά υπήρξαν μεγάλα ε, ζητήματα και θα ήθελα να μας πείτε και εσείς την δική σας αξιολόγηση. Κατά δεύτερον, πιστεύω ότι οι εθνικέ μονάδε μυστικών υπηρεσιών σε κεντρική, με κεντρική διαμόρφωση συχνά δεν αφήνουν να συμμετάσχει όσο πρέπει η αστυνομία και οι δυνάμει ασφαλεία. Και από πλευρά τη Europol διαπιστώθηκε, για παράδειγμα, στη Γαλλία ότι υπάρχει ανάγκη να συμμετάσχει πολύ πιο πολλέ στι δράσει και η περιφερειακή αστυνομία, γιατί αυτοί είναι εκείνοι που βλέπουν στην πρώτη γραμμή αν θέλετε, στο πρώτο επίπεδο τι συμβαίνει. Γιατί υπάρχουν πολλά συμπτώματα τα οποία δεν είναι αρκετά εντυπωσιακά, αν θέλετε, για να κοινοποιηθούν στις εθνικές αρχές ασφάλειας. Θα πρέπει υπάρχει, για παράδειγμα, προσβασιμότητα στο σύστημα ΣΕΝΑ. ένα η προσβασιμότητα στην παρούσα φάση είναι πάρα πολύ περιορισμένα γιατί το σύστημα ΣΕΝΑ έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο που η άμεση πρόσβαση στο σύστημα δεν επιτρέπεται ουσιαστικά σε τοπικούς φορείς. Τελευταία ερώτηση για το θέμα της κινητοποίησης των μουσουλμάνων. Μας είπατε για αυτά τα 56.000 άτομα, από τα οποία 10.000 είναι πραγματικά επικίνδυνα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που δεν ενδιαφέρει όλους ιδιαίτερως είναι το εξή. όλο αυτό το οικοσύστημα. Τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, όπως τα κατανοούμε εμείς, κράτος δικαίου, ισότητα των φύλων, ανεξιθρησκεία, όλες αυτές οι αρχές λοιπόν. Πώς μεταφέρονται στα άτομα αυτά τα οποία έρχονται σε μας ε, ή μένουν μαζί μας ως μουσουλμάνοι, προκειμένου αυτό να καταστεί ένα κοινό σύστημα αξιών, είτε είναι χριστιανοί, βουδιστές, ε, ανεξαρτήτως θρησκείως. Θα πρέπει λοιπόν αυτά τα βασικά θεμελιώδη δικαιώματα να είναι οι ύψιστοι, οι ύψιστες αξίες και κοιτώντας τις δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει τελευταία δημοσκόπηση και από το Βέλγιο και από τη Γερμανία και τη Γαλλία σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την ισότητα ε, των φύλων. Συχνά η απάντηση είναι αρνητική. Όχι. Ή σε τελική ανάλυση ποιος ε, είναι αυτός που θα κρίνει μια διαφορά. 99% στις κοινότητες αυτές οι απάντησεις είναι ο ημάμις και όχι ε, ο δικαστής. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε πώς μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα κοινό σύστημα αξιών, γιατί το οικοσύστημα της δημοκρατίας μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν ο κόσμος αμφιβάλλει για τις αξίες αυτές. Όταν οι αξίες είναι σαφές δεν υπάρχει και καμία αμφιβολία. Αν θα μπορούσατε λοιπόν να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω από αυτού Πολλές ερωτήσεις, ε, πολλές και διαφορετικές, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Θα, θα προσπαθήσω να απαντήσω. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση, τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση οι τρομοκράτες σε πυρηνικά, βιολογικά, χημικά προϊόντα και το καθεξής. Αυτό που με ανησυχεί είναι η πιθανή πρόσβαση ε, των τρομοκρατών στις πρόδρομες ουσίες για την κατασκευή εκρηκτικών υλικών. Και μάλιστα και πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν εφαρμόσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία, την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, ώστε όταν κάποιος πάει να αγοράσει ένα προϊόν που είναι πρόδρομη ουσία για εκρηκτικά, καταγράφεται το όνομά του, τα στοιχεία του. Πολύ καλό αυτό. Αλλά η σχετική νομοθεσία ισχύει στη θεωρία. Ε, και στον πραγματικό κόσμο. Τι γίνεται όμως με το διαδίκτυο, με τον εικονικό κόσμο. Εκεί μπορεί κάλλιστα να αγοράσει κανείς ανώνυμα ε, εκρηκτικά ή ε, πρόδρομες για τα εκρηκτικά και για το διαδίκτυο. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο μητρό που να καταγράφονται οι αγοραστές. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιώσουν τα πράγματα και στο διαδίκτυο, στην εικονική πραγματικότητα. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η εικονική πραγματικότητα. Και αυτή είναι η μορφή μας προς τους η κριτική μας προς τους νομοθέτες, που ναι μεν ακολουθούν τη δική τους λογική, μερικές φορές όμως αυτή είναι αποσυνδεμένη από την ε, πραγματικότητα που είναι πιο σφαιρική και έχει και εικονική διάσταση. Τώρα, για ε, την ε, εμπλοκή των τοπικών παραγόντων, αστυνομικών και ούτω καθεξής. Το θέμα είναι περίπλοκο το φαινόμενο και η, ριζ, ριζοσπαστικοποίηση δεν αφορούν την αστυνόμευση. Είναι ιδεολογικό το θέμα. Αν έχουμε την παραμικρή πόνοια για την συμμετοχή κάποιου σε δημοκρατικές οργανώσεις, τότε μπορούμε να ασκήσουμε δίωξη, να γίνει προσωρινή κράτηση. Αυτό είναι εύκολο. Το ιδεολογικό ζήτημα είναι πολύ πιο δύσκολο. Το θέμα της αστυνόμευσης είναι πιο εύκολο και συγκεκριμένο και θα πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ των κεντρικών αρχών του κράτους και ε, των φορέων που πιο εύκολα θα εντοπίσουν τα φαινόμενα της ριζοσπαστικοποίησης. Δεν είναι μόνο θέμα αστυνομικό ή αστυνόμευσης. Και μάλιστα ο συντονισμός των μονάδων των αντιτρομοκρατικών γίνεται στη Γαλλία με ένα νέο σύστημα που προβλέπει μεγαλύτερο συντονισμό και μία συγχώνευση μερικές φορές των διαφόρων αντιτρομοκρατικών ομάδων. Και μάλιστα σκεφτήκαμε να το γενικεύσουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί ο κίνδυνος είναι εξορισμού διασυνοριακός. Γιατί πρόκειται για πρόσωπα που, και άτομα που περνάνε τα εθνικά σύνορα. Και να μην ξεχνούμε ότι το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα περιθωριακό. Η μεγάλη πλειοψηφία των μουσουλμάνων στις χώρες μας ε, προσ... το σύστημα αξιών μας, των δημοκρατικών μας αξιών πλήρως. Μιλούμε για ε, ένα ελάχιστο τμήμα των μουσουλμάνων που το αφισβητούν. Πρόκειται για περιθωριακούς ε, μουσουλμάνους που έχουν κάποιες διεκδικήσεις και ιδεολογικές και θρησκευτικές που δεν έχουν καμία σχέση, δεν έχουν κανένα κοινό σημείο με την συντριπτική πλειοψηφία των υπόλοιπων μουσουλμάνων. Οπότε δεν θα πρέπει να τους ηχαίουμε που δεν είναι. Το πρόβλημα δεν είναι οι μουσουλμάνοι απέναντι στις δημοκρατικές αξίες, αλλά το πρόβλημα συγκεκριμένων ατόμων με ιδεολογικές πολιτικές ε, βλέψεις και διεκδικήσεις, που είναι μια εξαιρετικά μικρή μειοψηφία των μουσουλμάνων, ένα περιθωριακό τμήμα. Και φυσικά θα πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε διαφυλάσσοντας ε, τις δημοκρατικές μας ε, αξίες. Ευχαριστώ. Η Χέλγα Στίβεν τώρα, η δεύτερη μα εισηγήτρια, ή μάλλον συνεισηγήτρια, γιατί πρώτο και δεύτερο δεν υπάρχει, είναι συνεισηγήτρια ισότιμε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλου. Σα Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήλθατε, κύριε Μπριτσάρ. Δυστυχώς διαπιστώνω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σα. Το 2018 στην καταπολέμηση τη τρομοκρατία ε, δεν έχουμε ακόμα κάνει τα σημαντικά βήματα που θα πρέπει να έχουμε κάνει. Αντιμετωπίζουμε σημαντικέ προκλήσει και μία από τι προκλήσεις αυτές είναι η διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, η οποία παραμένει σημαντικό ακαθόδες σημείο, τουλάχιστον οκτώ από τους υπέτειους στις επιτέσεις του Παρισιού ήταν Σύριοι, οι οποίοι είχαν επανέλθει εκεί μέσω από τον νησί της Λέρου στην ε, ε, Ελλάδα και από ουγγρικά εδάφη και ε, έκαναν ότι είναι πρόσφυγες. Ε, κύριε Μπριζάρ, ε, με τις γνώσεις σας και με την εμπειρία σας ήθελα να σας ρωτήσω τι πιστεύετε ότι δεν προσέχουμε παρκώς. Μπορείτε να μας πείτε τι κενά πιστεύετε ότι υπάρχουν ακόμα στην ε, διασφάλιση των εξωτερικών μας συνόρων και μήπως έχετε κάποιες συστάσεις να κάνετε τις οποίες θα, συμπεριλάβουμε στην έκθεσή μας. Ευχαριστώ πολύ. Merci bien. Ευχαριστούμε την Έλγα. Ευχαριστώ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, λέει ο κ. Μπρίσαρ. Το κέντρο ανάλυσης του οποίου προεδρεύω ασχολείται ακριβώς με, αυτό, ασχολείται ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Με τον τρόπο δηλαδή που επιστρέφουν οι τζιχαντιστές μέσω των μεταναστευτικών οδών των Βαλκανίων. Το 2015 μέσω της Σερβίας, μέσω της Μακεδονίας, είχαμε καταγράψει, της Ουγγαρίες είχαμε καταγράψει τέτοια περιστατικά, καταλήγουν στην Αυστρία ή στην Γερμανία. Είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα αυτό. Όπως ε, υπογραμμίσαμε, η Ευρώπη έχει κάνει προόδους, έχει τροποποιήσει τη συνθήκη του Σέγγεν. Αυτό που είναι σημαντικό για μας, για να μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα, είναι η τεχνικές των ίδιων των τρομοκρατών. Οι τρομοκράτες έχουν καταφέρει να προσαρμοστούν και να αναπτύξουν τις, τις δικές τους τεχνικές ώστε να μπορούν να παρισφρύνουν στις μεταναστευτικές ροές. Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ότι κάποια άτομα έχουν πρόσβαση, κάποιες τρομοκρατικές οργανώσεις έχουν πρόσβαση στην ε, Τουρκία από όπου μπορούν να προμηθεύονται πλαστά χαρτιά, πλαστά διαβατήρια και χάρη σε αυτά τα πλαστά διαβατήρια μπορούν να ταξιδέψουν, μπορούν να μπουν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ιδού λοιπόν ένας νέος τρόπος, ένας νέος δρόμος που επιτρέπει στους τρομοκράτες που θέλουν να επιστρέψουν, να χτυπήσουν ενδεχομένως στην Ευρώπη. Δεν θέλω να παρουσιάσω σε λεπτομέρειες, να επισέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά σε γενικές γραμμές αυτό το βλέπουμε τον τελευταίο καιρό. Θέλω να επιστρέψω στον τρόπο με τον οποίο οι τρομοκράτες εκμεταλλεύονται τις μεταναστευτικές ροές, τις μεταναστευτικές οδούς, έχουν μια παγκόσμια, θα λέγαμε, στρατηγική, διότι το χαλιφάτο έχει βεβαίως γεωγραφικά όρια εκεί όπου εδρεύει το Ισλαμικό κράτος. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι έχουν τροποποιήσει εντελώς τα μοντέλα επιθέσεων. Θέλουν να επιστρέφουν σε ευρωπαϊκό έδαφος με μονομένα άτομα, ούτω ώστε να μπορούν πολύ γρήγορα να χτυπούν. Τα άτομα αυτά έχουν ευρωπαϊκά διαβατήρια. Και περνάνε στη, στη θάση, περνάνε στην πράξη. Δεν είναι ιδιαίτερα εκπαιδευμένα, καλά εκπαιδευμένα τα άτομα αυτά. Έτσι υπάρχουν και αρκετές αποτυχίες. Αυτό συμβαίνει τον Ιούνιο του 2015 όταν ε, μια χώρα των Βαλκανίων αποφάσισε να ανοίξει τα σύνορά της. Είχαμε άτομα που εμπλέκονται στις επιθέσεις στις Βρυξέλλες και στο Παρίσι, πέρασαν τον έλεγχο των διαβατηρίων, εποφελήθηκαν λοιπόν αυτή τη ευκαιρία και το καλοκαίρι του 2015 κατάφεραν να περάσουν τα σύνορα. Πρόκειται για μια στρατηγική του Ισλαμικού κράτους. Ιδού η απάντηση. Ευχαριστούμε για τις διασαφηνίσεις από το 2015. Ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα καλυτερεύσουν. Δίνω το λόγο στον επόμενο ομιλητή. Ξεκινήσαμε λίγο αργά, έχουμε λίγη ακόμη ώρα. Δεν ξέρω αν πρέπει να φύγετε αμέσως, λέει η πρόεδρος. Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα μιλήσω ισπανικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι παρατηρήσεις σας και η παρέμβασή σας. Θα ήθελα να πω Να σας ευχαριστήσω για αυτά που μας είπατε, κοιτώντας και τα διάφορα μοντέλα χρηματοδότησης. Διαπιστώνουμε ότι ευτυχώς, ευτυχώς δεν έχουν τις ικανότητες που θα χρειάζονται για τη δημιουργία όπλων και όπλων μαζικής καταστροφής. Υπάρχει μια προσέγγιση χαμηλού κόστους, ευτυχώς. Αλλά αυτό που επισημάνεται είναι ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα και κάποιες ελλείψεις. Δεν μπορούμε να εντοπίσουμε καν κάποιους από τους πόρους που χρησιμοποιούνται σε ριζοσπαστικοποιημένες τέτοιες ε, μονάδες, ε, κοιτώντας τι γίνεται και στη Γαλλία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Νομίζω ότι οι υπόλοιπε χώρε πολλά μπορούν να διδαχτούν από τη Γαλλία. Έχετε πολλά να μα μάθετε. Μπορείτε να μα βοηθήσετε να κατανοήσουμε πώς θα μπορεί να διακοπεί αυτός ο φαύλος κύκλος και πώς μπορούμε να παρέμβουμε σε αυτό το σύστημα που έχει σχεδιαστεί ουσιαστικά για να μην μπορεί να εντοπίζεται. Στο σημείο λοιπόν αυτό θεωρώ ότι μπορούμε να υποφεληθούμε από την εμπειρία σας. Κοιτώντας λοιπόν τι έχετε κάνει και στην Γαλλία, έχετε εντοπίσει περιπτώσεις ε, τέτοιων περιπτώσεων, τέτοιων ε, τοξικών ατόμων, τοξικών ε, κοινοτήτων, όπου η ριζοσπαστικοποίηση έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο προκειμένου να υπάρχει απειλή για την κοινωνία. Και από την άλλη πλευρά θα ήθελα να μου πείτε αν έχετε εντοπίσει πολλές περιπτώσεις κοινοτήτων όπου θα ήταν δύσκολο να κάνουμε διάκριση μεταξύ του βίαιου φανατισμού από την θρησκευτική ριζοσπαστικοποίηση. Γιατί έχουν πολλά κοινά σημεία. Αυτοί που είναι θρησκευτικά φανατικοί και αυτόν που είναι βία φανατικοί. Ποια είναι η δική σας εμπειρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ε, καταρχήν, έχουμε πολλέ, πολύ επικάλυψη θρησκευτικής ε, και φανατικής ε, ριζοσπαστικοποίηση, βίαιης ριζοσπαστικοποίηση, ούτε υπάρχει ένα νέο προφίλ, ούτε ένα καλούπι. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιοι τρομοκράτες προέρχονταν από εγκληματικά κυκλώματα. Ήταν μικροεγκληματίες και είναι πολλοί αυτοί και δεν είναι κάτι το καινούριο. Εδώ και καιρό είχαμε τέτοιο φαινόμενο που οι δύο κόσμοι της εγκληματικότητας και της ριζοσυσκοποίησης συμβαδίζουν και έχουν κάποιες ε, επαφές και επικαλύψεις. Και μερικές φορές ε, μια οργανωτική στήριξη των ριζοσπαστικοποιημένων προερχόταν από την οργανωμένη εγκληματικότητα. Σε ό,τι αφορά τα θέματα εκβιασμού ή μικρών υποθέσεων εκβιασμού και αφαίρεσης χρημάτων. Ε, δεν έχω υπόψη μου συγκεκριμένα θέματα στη Γαλλία ή στο Βέλγιο ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν μου έρχονται τουλάχιστον ε, έτσι αμέσως. Και να επανέλθω στο θέμα της μικροχρηματοδότησης. Ε, διαπιστώνουμε ότι οι τρομοκράτε για να οργανωθούν δεν χρειάζονται και πολλά χρήματα είτε για να, επιστρέψουν στις εμπόλεμες περιοχές ή να οργανώσουν μια τρομοκρατική επίθεση. Για θέματα εκβιασμού, για χρησιμοποίηση, για αποκομιδή χρημάτων δεν έχω συγκεκριμένες υποθέσεις και η κυρία Μπέρν είναι η τελευταία μας ομιλητρία. Θα μιλήσω σου ειδικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπριζέρ. Και θα ήθελα πάρα από αυτά που είπε η κυρία Στίβενς να προσθέσω και το εξή. Το 2015 και το 2016 ήταν μεγάλες ε, οι μεταναστευτικές ροές και ξέρουμε ότι μεγάλος αριθμός τρομοκρατών υπησύλλεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις, μεταναστευτικέ με ροέ. Ε, μεταναστευτικές αυτές ροές. Αναφερθήκατε στο θέμα του ελέγχου των συνόρων. αλλά από τις 12 Μαΐου και μετά δεν θα μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτόν τον έλεγχο στα σύνορά μας, εκτός και να αλλάξει κάτι στον κώδικα του Σέγγεν. Άρα υπάρχει αυτό το διακύβευμα να ξεκινήσουν καινούργιες μεταναστευτικές ροές και το έχει σκεφτεί κανείς αυτό, έχει σκεφτεί κανείς αυτή τη διάσταση της ε, ασφάλειας των σύνορων. Νέε προκλήσει επίση αναφέρατε. Εγώ θα έλεγα πιο πολύ νέε απειλέ. Βλέπω ότι υπάρχει απειλή όταν έρχεται κόσμο μαζικά, μαζικά τα τελευταία χρόνια και καταθέτει αίτηση για άσυλο παρά το γεγονό ότι δεν δικαιούται άσυλο, στην οποία περίπτωση φυσικά και διαφεύγουν και ζουν στην παρανομία, χωρίς χαρτιά. Για παράδειγμα, στην αγορά τη Χριστουγεννιάτικη στο Βερολίνο είδαμε ένα άτομο το οποίο ήταν χωρίς χαρτιά και στη Φιλανδία έγινε μία επίθεση από ένα άτομο το οποίο είχε απορριφθεί η αίτησή του για άσυλο. Πώς ε, λοιπόν θα τα καταφέρουμε και θα τα επεξελθούμε και στις προκλήσεις αυτές, στις απειλές αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Euh, για την ερώτηση αυτή. Κάθε χώρα, να σας πω, ότι κάθε χώρα έχει τη δική της πολιτική σε ό,τι αφορά τους, τους τη. της. Και ξέρω ότι σε διάφορες χώρες ε, οι αιτούντες άσυλο ελέγχονται, παρακολουθούνται από τις μυστικές υπηρεσίες ε, της χώρας και σε διάφορες περιπτώσεις ε, έχει γίνει σύνδεση και με κλιματικές ή τρομοκρατικές δραστηριότητες και έχουν καταδικαστεί. Κάθε λοιπόν ευρωπαϊκό κράτος έχει δική του πολιτική στο θέμα αυτό δεν βλέπω να υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή πολιτική πραγματικά σε αυτό το επίπεδο. Επανέρχομαι σε αυτό που είπα προηγουμένως, ότι οι δρομοκράτες ε, χρησιμοποιούν ε, αυτό το κενό σε ό,τι αφορά το κενό που υπάρχει στον έλεγχο του σύνορων, σε ό,τι αφορά το θέμα των Βαλκανίων το 2015, το είπαμε, ήταν προσωρινό φαινόμενο. Και έτσι εισήλθαν ε, στα σύνορα αυτά, στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, τρομοκράτες, ε, άτομα τα οποία πέρασαν με πλαστά έγγραφα κτλ. Ήταν μια συγκεκριμένη περίπτωση όπου διαπιστώθηκαν κενά στα αμυντικά μας συστήματα και ήμασταν ανήμποροι απέναντι στην αναχέτηση των τον τρομοκρατών να εισέλθουν στο έδαφος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπριζάρ. Ευχαριστώ που είχατε την καλοσύνη να απαντήσετε στην πληθώρα των ερωτήσεων με πολύ σαφή και συγκεκριμένο τρόπο που θα μας βοηθήσει ιδιαίτερο και στην εκπόνηση της έκθεσής μας. Και σας ευχαριστώ για την ενέργεια, τη σαφήνεια, τη διάβγεια που χαρακτήρισαν την τις παρεμβάσεις σας. Χίλια ευχαριστώ εκ μέρους των μελών της Επιτροπής και σας ευχόμαι και καλή επάνωδο στο Παρίσι. Καλό ταξίδι. de changement. Ah, c'est bon. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ να καθίσετε στη θέση σας. Περνάμε στο δεύτερο σημείο, την ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Ραφαήλ Μαλανινή, τον ε, η εισαγγελέα, ομοσπονδιακό δικαστή, θα μας μιλήσει για την συνεργασία στην καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Όπως γνωρίζετε, τα μέτρα που έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν συμμορφωθεί με τις συστάσεις του ΓΚΑΦΗ, της ομάδας χρηματικών υποθέσεων, και βέβαια σύμφωνα με το Συμβούλιο Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών. Σε αυτές τις συστάσεις, τις ειδικέ συστάσεις, όλες οι χώρες α, θα πρέπει να συνεργάζονται σε νομικό πλαίσιο, σε ό,τι αφορά τις έρευνες, σε ό,τι αφορά τις ποινικέ διώξεις, σε ό,τι αφορά τα διοικητικά ζητήματα που αφορούν στην ε, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Σε ενωσιακό επίπεδο τώρα η νομοθεσία που αφορά το ξέπλυμα του χρήματος, την, ε, κυκλοφορία, την παράνομη κυκλοφορία μετρητών ε, και το πάγωμα αλλά και τις κατασχέσεις. Το σχέδιο δράσης της Κομισιόν του 2 Φεβρουαρίου του 2016 βασίζεται κυρίως στην πρόληψη αλλά και στον εντοπισμό που βασίζεται στη λογική follow the money, ας ακολουθήσουμε τα χρήματα δηλαδή, γιατί το να μπορούμε να εντοπίζουμε τις ε, χρηματοοικονομικές, ε, ύποπτες χρηματοοικονομικές ροές μας επιτρέπει να μπορούμε να εντοπίζουμε και τους ίδιους τους τρομοκράτες. Αυτό το σχέδιο δράσης λοιπόν αφορά στην ενδυνάμωση των αρμοδιοτήτων των πυρήνων πληροφορίας, οικονομικών πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στο να δευκολύνει την συνεργασία μεταξύ των διαφόρων αυτών κέντρων πληροφοριών, ούτως ώστε να μπορέσουμε να εξαλείψουμε την, το ξέπλυμα του, του χρήματος. Κύριε Μαλανίνη, η εμπειρία σας σε ό,τι αφορά την νομική συνεργασία στην αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Επιτροπή μας, ε, ιδίως για τις συνσυνηγήτριες. Και αν είστε λοιπόν σύμφωνοι, ε, θα ήθελα να σας προτείνω να πάρετε το, το λόγο για 20 λεπτά και στη συνέχεια αν είστε σύμφωνος να απαντάτε με τη μέθοδο αυτή ping-pong. Θέλω λοιπόν να σας προτείνω, λέει ο κύριος Μαλανίνη, στα 20 λεπτά που θα μιλήσω μία ανάλυση του, του πεδίου. Τι προκύπτει λοιπόν σε νομικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Θέλω λοιπόν πρώτα απ' όλα να θίξω το ζήτημα που έχει να κάνει με τους περιορισμούς της νομοθεσίας έτσι ως έχει. Να μιλήσουμε λίγο για το ευρωπαϊκό δίκαιο και γιατί τα μέτρα που έχουμε λάβει είναι κυρίως ευρωπαϊκά. Το δεύτερο ζήτημα που θέλω να ζήξω στην παρουσίασή μου είναι ότι παρά τους περιορισμούς του είναι αρκετά χρήσιμο το σύστημα που χρησιμοποιούμε. Θα σας το παρουσιάσω αυτό με δύο παραδείγματα. Το τρίτο σημείο έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση των λεγόμενων foreign terrorist fighters, των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών. Και εδώ η συνεργασία, η νομική συνεργασία και η συνεργασία της αστυνομίας στην Ευρώπη είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Σε ό,τι αφορά Θέλω να σας δώσω και ένα παράδειγμα για τη συνεργασία μεταξύ Γαλλίας και Βελγίου, ακριβώς αυτό το σημείο συνεργασίας καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Το ζήτημα αυτό είναι ένα ζήτημα αντίδρασης που αφορά βεβαίως σε γενικές γραμμές το φάκελο τρομοκρατία και θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην καταπολέμηση των τρομοκρατικών χτυμάτων γενικά. Θέλω να ξεκινήσω λοιπόν η... λέγοντας ότι η καταπολέμηση της χρηματοδότησης της θερμοκρατίας ξεκινάει ουσιαστικά το 2001 μετά την μετά τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001. Α, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις 28 Σεπτεμβρίου του 2001 ζητά να καταπολεμηθεί η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και να ποινικοποιηθεί. Οι αρχές αυτές της 28 Σεπτεμβρίου του 2001, το ψήφισμα αυτό, ίσως ξεκινήσαμε λίγο με λάθος βάση. Υπό τη ότι οι τρομοκρατικές οργανώσεις, θεωρώντας ότι οι τρομοκρατικές οργανώσεις έχουν ανάγκη από πολλά χρήματα προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις επιθέσεις τους και ότι χρησιμοποιούν τις συμβατικές τραπεζικές οδούς. Η αλήθεια όμως είναι ότι οι πολύ νεκρές τρομοκρατικές επιθέσεις συχνά έχουν πολύ χαμηλό κόστος. Πράγμα που δεν σημαίνει βεβαίως ότι οι τρομοκρατικές οργανώσεις δεν έχουν ανάγκη από χρήματα. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια α, ασυμμετρία σε ό,τι αφορά τα χρήματα που χρησιμοποιούνται για να πραγματοποιηθεί μια τρομοκρατική επίθεση και το κόστος που έχουν για τα άτομα που θα έχουν υποστεί την επίθεση οι εκτιμήσεις που αφορούν την 11η Σεπτεμβρίου, για παράδειγμα, οι τρομοκράτες επένδυσαν ε, περίπου 200 με 500 χιλιάδες δολάρια και το κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες ανέρχεται στα χίλια δισεκατομμύρια δολάρια. Όπως βλέπετε υπάρχει μια τεράστια απόσταση ανάμεσα στα χρήματα που εντός αγωγικών επενδύθηκαν και στη ζημιά που η τρομοκρατική επίθεση αυτή επέφερε. Βεβαίως, το γεγονός ότι οι τρομοκρατικές οργανώσεις δεν έχουν ανάγκη από χρήματα είναι ένας αστικός μύθος. Βεβαίως και έχουν ανάγκη από χρήματα για να χρηματοδοτήσουν την οργάνωσή τους, για να μπορέσουν να διοχετεύσουν την προπαγάνδα τους και να πληρώσουν τους μαχητές τους. Το έχουμε δει στην περίπτωση του ΠΚΚ, όπου χρησιμοποιεί περίπου 80% των πόρων του για να μπορέσει να αδιοχετεύσει την προπαγάνδα του. Σε επίπεδο ε, των περιορισμών τώρα της υπάρχουσας νομοθεσίας, θέλω να αναφέρω ένα άρθρο του Peter Newman, δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2017. Το άρθρο αυτό έχει τον τίτλο Don't follow the money, κάνοντας ένα λογοπαίγνιο με την αρχή του Bush follow the money που αναφέραμε νωρίτερα. Το Ισλαμικό κράτος σύμφωνα με τον Νιούμαν, είχε έναν προϋπολογισμό της τάξης του 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2015 και τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν παγώσει αντιστοιχούσε σε περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια το 2015. Βλέπετε λοιπόν ποια είναι η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα χρήματα που είχαν στη διάθεσή τους οι τρομοκράτες και στα χρήματα που είχαν ε, παγώσει ως αποτέλεσμα των μέτρων της καταπολέμησης χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. σύμφωνα με τον συγγραφέα είναι μάταιο να προσπαθούμε να σταματήσουμε την χρηματοδότηση της ε, τρομοκρατίας ε, παρακολουθώντας το χρηματοοικονομικό σύστημα. Γιατί δεν χρησιμοποιούν απλούστατα τα συμβατικά τραπεζικά κυκλώματα οι τρομοκράτες. Μάλιστα ο συντάκτης του άρθρου επισήμανε και ένα αντιπαραγωγικό στοιχείο. Οι οργανισμοί μεταφοράς χρημάτων δεν συνεργάζονται με κάποιες επικίνδυνες χώρες όπως την Σομαλία για παράδειγμα. Και επίσης τέτοιοι οργανισμοί αρνήθηκαν να συνεργαστούν με τη Σομαλία ενώ υπήρξαν τεράστια προβλήματα στη Σομαλία, γιατί περίπου 40% του πληθυσμού εξαρτώνταν από εμβάσματα που προέρχονταν από την Αλοδαπή, από χρήματα από το εξωτερικό και τέτοιες μεταφορές αποστολές μάλλον χρημάτων σε ό,τι αφορά του πόρου του Ισλαμικού κράτου και τη χρηματοδότηση. Αυτό δεν γίνεται από τα κλασικά τραπεζικά κυκλώματα, αλλά από τα εδάφη που ελέγχει το Ισλαμικό κράτος, από τη δίμευση των περιουσιακών αγαθών των κατοίκων, από την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων του ελεγχόμενου ε, της ελεγχόμενης επικράτειας και στο μέτρο που η οργάνωση αυτή μετατρέπεται σχεδόν σε ιονή κράτος, ε, αρχίζει και δημιουργεί και έξοδα, θα έχει έξοδα για το διδακτικό προσωπικό, για το δικαστικό σύστημα που σύστησε, έξοδα της γραφειοκρατίας και έξοδα που είναι επακόλουθα της δημιουργίας ενός ιονή κράτους. Και μάλιστα οι τρόποι χρηματοδότησης ε, εκφεύγουν ε, του ελέγχου και της επιτήρησης ε, των δικαστικών αρχών βελγικών ή άλλων. Δεν γνωρίζω κανέναν δικαστή που να γνωρίζει τι συνέβη, πώς έγινε η χρηματοδότηση του Ισλαμικού κράτους στη Συρία ή το Ιράκ. Αυτή η χρηματοδότηση του Ισλαμικού κράτους μέσω του Σύρο-Ιρακινής ζώνης ουσιαστικά παρεμποδίστηκε από άλλα μέτρα για παράδειγμα το εμπάργο που αποφασίστηκε σε διεθνές επίπεδο και κάποιες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, σε ένα άρθρο του Νόιμαν αναφέρει το παράδειγμα ενός ε, αμερικανικού βομβαρδισμού που τον Ιανουάριο του 2016 ε, καταστρέφει ε, μία αποθήκη με δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά που είχε το Ισλαμικό κράτος. Οπότε έτσι όντως παρεμποδίστηκε χρηματοδότηση και μάλιστα με ε, πολύ πιο εντυπωσιακό τρόπο από ότι η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των τρομοκρατικών οργανώσεων που ήταν μόνο τη τάξη των 60 εκατομμύριων. και είχαμε καταστροφή δεκάδων εκατομμύριων. Πολύ περισσότερο. Τώρα, ε, για τη χρηματοδότηση των τρομοκρατικών επιθέσεων στην Ευρώπη. Νομίζω το ξέρετε ότι ο προπολογισμό του είναι πενιχρό και μάλιστα μία μελέτη του Ιανουαρίου του 2015 τη Εμιλίου Αφτεντάλ ναι, που μελέτησε 40 τρομοκρατικούς πυρήνες ε, από το 1994 με το 2013 και κατέληξε ότι ο μέσος προϋπολογισμός τους είναι περίπου 10.000 δολάρια. Η μελέτη αυτή καθορίζει ότι τα μέτρα χρηματοδο... μέσα χρηματοδότηση της τρομοκρατίας είναι κυρίως προσωπικά. 58% των του πόσου που χρειάζεται για τη διάπραξη μιας τρομοκρατικής επίθεσης προέρχεται από τον ίδιο τον τρομοκρατικό πυρήνα. Ένα στους τέσσερις πυρήνες μόνο έχουν λάβει χρηματοοικονομική υποστήριξη από την τρομοκρατική οργάνωση που διεκδίκησε την τρομοκρατική επίθεση. Ουσιαστικά δηλαδή περισσότεροι τρομοκρατικοί πυρήνες αυτοχρηματοδοτούνται. Οπότε θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας για να εντοπίσουμε και να αποτρέψουμε κάποιες τρομοκρατικές επιθέσεις, δεν θα τα καταφέρουμε. Ακριβώς γιατί δεν ακολουθούν αυτά τα κυκλώματα. Επίσης, τα οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη επιβεβαίωσαν τη διαπίστωση του ισχυρού προπολογισμού. Το... Στο Παρίσι στις 13 Νοεμβρίου 2015 Μα δείχνει μία μελέτη του κυρίου Μπριζάρ ότι ο προπολογισμό που χρειάστηκε ήταν 82.000 ευρώ για τι τρομοκρατικέ επιθέσει του Παρισιού τη 13 η Νοεμβρίου 2015. Οπότε μιλούμε πολύ χα... Ε, σε άλλε περιπτώσει για πολύ χαμηλότερα ακόμη κονδύλια. Για παράδειγμα, στι 14 Ιουλίου του 2016, στην τρομοκρατική επίθεση τη Νίκαια, ε, που οδήγησε στο θάνατο 86 ανθρώπων, ουσιαστικά το κόστο τη τρομοκρατική επίθεση ήταν η ενοικίαση τη Δαλίκα. Ενώ στο Βερολίνο το Δεκέμβριο του 2016 που είχαμε αντίστοιχη ε, επίθεση με Νταλίκα σε χριστουγεννιάτικη αγορά με 12 νεκρούς. Εκεί ήταν τελείως ανέξοδη η οργάνωση γιατί ο δράστης έκλεψε την Νταλίκα και την ε, έριξε πάνω στο κοινό. Επίσης στο Βέλγιο, στο, ε, στην τρομοκρατική πίεση του Σερλερό 6 Αυγούστου 2016 είχαμε σοβαρό τραυματισμό δύο αστυνομικών με μαχαίρι που δανείστηκε από φίλο του. Επίσης, στις 20 Ιουνίου του 2017, στο σταθμό, συντεροδομικό σταθμό των Βρυξελών, κάποιος προσπάθησε να ανατιναχθεί στη, στο, σιδηροδρομικό σταθμό. Ευτυχώ ε, δεν λειτουργήσε ο μηχανισμό. Εκεί χρειάστηκα μερικά, μερικά εκατοντάδε ευρώ για να αγοράσει μια βαλίτσα, ε, μια φιάλη αερίου και βίδε, ε, παξιμάδια για να δημιουργήσει αυτόν τον εκρηκτικό μηχανισμό και μάλιστα ήταν πολύ εύκολο να προμηθευτεί οπουδήποτε αυτά τα υλικά. Χαμηλότατο ο προπολογισμό λοιπόν. Όλα αυτά για να σα αποδείξω ότι κατά τη γνώμη μου τα μέτρα χρηματοδότηση ή μάλλον πολέμηση τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία ε, έχουν πολύ περιορισμένο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την ισχύουσα, την παρούσα τρομοκρατική απειλή και την ε, αποτροπή τρομοκρατικών επιθέσεων ή την πρόληψη σε τέτοια θέματα. Δεν θα έλεγα βέβαια ότι είναι τελείω άχρηστα αυτά τα μέτρα, επουδενή. Και μάλιστα θα σας δώσω δύο παραδείγματα που δείχνουν ότι τα μέτρα καταπολέμησης της χρηματοδότησης τρομοκρατίας ήταν αποτελεσματικά. Το ποινικό δικαστήριο των Βρυξελών ε, στις 21 Μαρτίου 2013 είναι απλέ υποθέσει διεθνού συνεργασίε, Οι ε, γαλλικέ αρχέ ενημερώνουν τι βελγικέ αρχέ για το ότι δύο Λιβανέζοι θα εμφανιστούν στο αεροδρόμιο Ζάβεντεμ για να πάρουν αεροπλάνο για το Λίβανο και καλό θα ήταν να ελεγχθούν οι αποσκευέ του. Έτσι και έγινε και στι αποσκευέ του βρέθηκαν μετρητά περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ και κάτι ψηλά και μάλιστα δεν μπόρεσαν να εξηγήσουν την προέλευση αυτού του πακτόλου. Μάλιστα ε, με την υπόθεση αυτή δεν ε, αποδείχθηκε η διασύνδεσή τους με τρομοκρατική οργάνωση. Οπότε όλες οι παραβάσεις σε σχέση με χρηματοδότηση τρομοκρατίας δεν ενεργοποιήθηκαν. Παρόλο που υπήρχαν σοβαρές υποψίες ότι είχαν τέτοια διασύνδεση με τρομοκρατική οργάνωση, αλλά δεν μπορούσαμε να το αποδείξουμε. Οπότε, ε, χάρη στι διατάξει για την καταπολέμηση τη νομοποίηση εσόδων από παράνομε δραστηριότητε ε, διώχθηκαν και καταδικάστηκαν σε τριετή φυλάκιση οι δύο αυτοί οι Λιβανέζοι και κατασχέθηκαν, ε, κατασχέθηκε το 1 εκατομμύριο ευρώ που μάλλον θα χρηματοδοτούσε τρομοκρατική οργάνωση. Χάρη λοιπόν στι ε, διατάξει για το ξέπλυμα χρήματο και μάλιστα το βασιλικό διάταγμα της 5ης Οκτωβρίου του 2006 ε, για τέτοια θέματα που εφαρμόστηκε την εκτέλεση σχετική νομοθεσία χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση αυτή για την καταπολέμηση της χρηματοδότηση τρομοκρατίας. Φαντάζομαι ότι αυτό ήταν ο πραγματικός λόγος, αν και νομικά ε, στοιχειοθετήθηκε το έγκλημα της, του ξεπλήματος χρήματος. Επίσης, ε, το Νοέμβριο του 2012 οι βελγικές ε, μυστικές υπηρεσίε, ενημερώνουν τις βελγικές δικαστικέ αρχές για τη συγκέντρωση κονδυλίων που έκαναν δύο άτομα ε, προ όφελο τη ε, κουρδική οργάνωση ΠΚΚ και μάλιστα βρέθηκαν μετρητά πάνω από 300.000 ευρώ μετά από τον έρωνο που έγινε υπέρ του ΠΚΚ. Επιλήφθηκε το ποινικό δικαστήριο τη Λιέγης. Οι άνθρωποι αυτοί διώχθηκαν με το κατηγορητήριο τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία με βάση το άρθρο 140 του ε, ποινικού κώδικα, γιατί έκαναν ένα είδος εκστρατείας καμπάνια, όπως το λέμε, που ήταν η επιβολή ενός είδους φόρου που αποφάζει η οργάνωση ΠΚΚ να επιβάλλει στους απόδημους ε, Κούρδους που ε, θέλοντας και μία έπρεπε να καταβάλουν το 10% των ετήσιων εσόδων τους στην οργάνωση ΠΚΚ. Επαναλαμβάνω, θέλοντας και εμεί το έκαναν, μερικοί και ο θελός και όλα. Ε, βέβαια υπήρξαν διαφωνίες για το κατά πόσο θα πρέπει να χαρακτηριστεί η οργάνωση ΠΚΚ ως τρομοκρατική και παρόλο που το αρμόδιο ποινικό δικαστήριο έγινε ότι δεν είναι τρομοκρατική η οργάνωση, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε εύλογο ότι ε, μια και τα δύο άτομα δεν ε, μπόρεσαν να δικαιολογήσουν την προέλευση των κονδυλίων αυτών, κατηγορήθηκαν τελικά για ξέπλυμα χρήματο για νομοποίηση εσόδων από παράνομε δραστηριότητε. Ιδού και το δεύτερο παράδειγμα τη ε, λειτουργικότητα των νομοθετικών διατάξεων και των δυνατοτήτων που μα ε, δίνουν για να καταπολεμήσουμε τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατίας. Και επανέρχομαι τώρα στην καταπολέμηση της χρηματοδότησης των ξένων μαχητών, τρομοκρατών μαχητών. Ε, πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες μετέβησαν στην Σύρο-Ιρακινή ζώνη και προσχώρησαν στην τρομοκρατική οργάνωση του Ισλαμικού κράτους. 400 είναι περίπου οι Βέλγοι ε, υπήκοοι που μετέβησαν στη Συρία ή το Ιράκ. Και μάλιστα χρηματοδότησαν το ταξίδι και τη διαμονή τους ε, κυρίως με δικούς τους πόρους, πολύ συχνά και με κοινωνικά επιδόματα Μάλιστα πολλοί ήταν άνεργοι και έλαβαν επίδομα ανεργία. Και μάλιστα από τη στιγμή της αναχώρησής τους μέχρι την διακοπή της χορήγησης του κοινωνικού επιδόματος ε, μεσολάβησε μεγάλο διάστημα και αυτά τα χρήματα ουσιαστικά ε, πήγαιναν μέσω του τραπεζικού του λογαριασμού στα άτομα αυτά. Οπότε το πρώτο μέτρο για την καταπολέμηση χρηματοδότηση τριμοκρατία σε βελγικό επίπεδο, όταν αντιμετωπίσαμε αυτό το θέμα των ξένων μαχητών, ήταν το συντομότερο δυνατόν να διακόψουμε την ε, καταβολή κοινωνικών επιδομάτων που χορηγούνταν στα άτομα αυτά. Από πληροφορίες που λάβαμε, ε, το Ισλαμικό κράτος ε, αντάμιβε τους ξένους μαχητές που στρατολογούσε. Βέβαια, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και τα μέτρα αποκλεισμού, εμπορικού αποκλεισμού του εμπάργου ουσιαστικά εξάντλησαν, τις, στέγνωσαν τις ε, οικονομικές πηγές του Ισλαμικού κράτους, οπότε έμειναν οι μαχητές αυτές ε, χωρίς, ε, οι μαχητές αυτές χωρίς χρήματα για την συντήρηση, την επιβίωσή τους, οπότε έστειλαν έκκληση βοηθείας προς τις οικογένειές τους, τους φίλους τους και τους ζήτησαν χρήματα για να συντηρηθούν ή να τους στείλουν τα επιδόματα ενεργείας ή τα άλλα κοινωνικά επιδόματα που είχαν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Όταν ενημερωθήκαμε για το φαινόμενο αυτό, δηλαδή ότι οι Βέλγοι επίκοοι έστειλαν, εμβάσματα ε, σε ξένους ε, τρομοκράτες μαχητές, FTF όπως τους λέμε, θεσπίσαμε διάφορους μηχανισμούς. Συνεργασία της Ευρωπόλ και των διαφορών οργανισμών ε, αποστολής χρημάτων. Έτσι εντοπίσαμε κάποια κυκλώματα χρηματοδότησης των ξένων μαχητών. Και μάλιστα χαρακτηρίσαμε αυτό το θέμα ως το συριακό πορτοφόλι. Αυτή ήταν συγκεκριμένοι που συγκέντρωναν τα χρήματα αυτά και τα έστεναν στη Συρία. Και μάλιστα όταν τα χρήματα αυτά φτάνουν προς Βέλγους που έχουν στρατευτεί στη Συρία, συνήθως χρησιμοποιείται η οργάνωση Western Union, μια οργάνωση αποστολής χρημάτων. Τα χρήματα αυτά στέλνονται από το Βέλγιο σε έναν αρμόδιο συγκέντρωσης συλλέκτικων δουλειών όπως το λέμε, ε, που βρίσκεται στο Λίβανο ή τη Συρία και μετά αυτός τα στέλνει στον, μαχητή του Ισλαμικού κράτους, ε, όπου και αν βρίσκεται. Και μάλιστα σε τέτοια περίπτωση βλέπουμε ότι ο ξένος μαχητής μέσω του WhatsApp ή άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μέσω του Ιντερνετ στέλνει το αίτημα στο Βέλγο και ε, λέει ποια στιγμή θα πρέπει να στείλει το έμβασμα και σε ποιον να στείλει αυτό το έμβασμα, ή στην Τουρκία ή στο Λίβανο. Και από τη στιγμή που φτάσουν τα χρήματα αυτά στην Τουρκία ή το Λίβανο, το Λίβανο μετά στέλνονται προς την Σύρο ηρακινη ζώνη ή μέσω ενός μηχανισμού αντιστάθμισης στυλ Αγουάλα ε, στέλνονται τα ευάσματα και βέβαια το Ισλαμικό κράτος λαμβάνει κάποια προμήθεια σε αυτή την αποστολή χρημάτων. Οπότε η αποστολή χρημάτων σε έναν μαχητή έμεσα χρηματοδοτεί και την τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό κράτο. Σε ό,τι αφορά τον εντοπισμό αυτών των επευθύνων συγκέντρωση των κονδύλων, των συλλεκτών κονδύλων, είναι εύκολο ο εντοπισμό του. Πρόκειται για του ίδιου του οργανισμού αποστολή χρημάτων που εντόπισαν αυτού του ε, συλλέκτε των κονδύλιων. Και είδαμε ότι κάποια ομάδα ανθρώπων λάβανε πολλά χρήματα χωρίς αποχρόντα λόγο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και μάλιστα από διαφορετικούς αποστολείς. Είχαμε δηλαδή έναν συλλέκτη κονδυλίων που μέσα σε λίγους εβδομάδες ή μήνες συγκέντρωνε ε, ποσά άνω των 80.000 ευρώ από διάφορες χώρες ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και εκτός αυτής, από το Καμερούν για παράδειγμα ή από άλλες χώρες. Οπότε δεν ήταν μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης λάβαμε αυτό το κατάλογο με τα άτομα αυτά που ε, συλλέκτες κονδύλιων και μετά κάθε εθνική αρχή είδε ποιοι υπηκοοί της έστελναν χρήματα σε τέτοιους ε, ε, συλλέκτες χρημάτων. Κατόπιν εξετάζαμε τον κατάλογο των Βέλγων στην περίπτωση του Βελγίου. Βλέπουμε Ποιο από το Βέλγιο έστενε χρήματα σε αυτόν τον συλλέκτη χρημάτων, κονδυλίων και ποιος, που έστελνε εκείνος τα χρήματα που συγκέντρωνε. Και έτσι μπορέσαμε να εντοπίσουμε ολόκληρο το κύκλωμα τέτοιων ε, συλλεκτών κονδυλίων και εντοπίσαμε και τους Βέλγους που έστελναν σε αυτούς τα κονδύλια. Η ανάλυση που έκανε το Τμήμα Οικονομικών Πληροφοριών του Βελγίου βοήθησε σε αυτό το θέμα, γιατί αυτό το τμήμα ανάλυση οικονομικών πληροφοριών ε, έδινε στην εισαγγελική αρχή τα στοιχεία ταυτότητας ε, των ε, δραστών αυτού του, του συριακού πορτοφολίου, αυτού του συλλεκτών κονδυλίων και έτσι ξεκινήσαμε πολλές δικαστικές υποθέσεις προκειμένου να αναχαιτήσουμε την χρηματοδότηση μεμονωμένων τρομοκρατών. Σε ό,τι αφορά τις ποινές, στην πρώτη δικαστική απόφαση της 26 Φεβρουαρίου 2018 από το ποινικό δικαστήριο του Ντάντερ Μόντε, η μητέρα και η αδερφή ενός μαχητή έστειλαν 10.000 ευρώ στον συγκεκριμένο τρομοκράτη μαχητή. Η έρευνα έδειξε ότι το ποσό αυτό το χρησιμοποίησε ο τρομοκράτης για να αγοράσει όπλο και η μητέρα του καταδικάστηκε σε 12 ε, μήνες φυλάκιση με αναστολή και η αδερφή τους 8 μήνες φυλάκιση. Επαναλαμβάνω, πρόκειται και ευρωπαϊκό ζήτημα και έχουμε και άλλε αποφάσει σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε που εκδόθηκαν για τέτοια θέματα. Για παράδειγμα, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο των Παρισίων ε, στι 28 Σεπτεμβρίου του 2017 ε, καταδίκασε σε διετή φυλάκιση τη μητέρα ενό τέτοιου μαχητή Μάλιστα στην Μεγάλη Βρετανία ήταν πολύ πιο αυστηρή η απόφαση γιατί για 219 λίρες τερλίνες που στάλθηκε από ένα θείο στον, στον τρομοκράτη ε, άνυψιό του καταδικάστηκε σε δύο χρόνια και τρεις μήνες φυλάκιση ο θείος. Επίσης στα κάτω χώρες η αποστολή χιλίων ευρώ ε, τιμωρήθηκε με 12 μήνη ε, φυλάκιση. Οπότε εφαρμόστηκε αστυνομική και δικαστική συνεργασία με μεγάλη επιτυχία κατά τη γνώμη μου στα πλαίσια αυτού του προβληματισμού της αναχέτησης χρηματοδότησης. Η Ευρωπόλ καταρχήν ερώθηκε από τη Western Junior και εξέδωσε τον κατάλογο με τους συλλέκτες των κονδυλίων ώστε να ασκήσουμε διάφορες ε, μηνύσεις και να ξεκινήσουμε διάφορες υποθέσεις. Επίση, η Eurojust επεσήμανε το ζήτημα αυτό στις δικαστικέ αρχές. Έγιναν σεμινάρια και συνεδριάσεις με κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων χωρών. Και η αρχή λειτουργία ήταν η απλούστατη. Κάθε χώρα θα διώκει τους υπηκόους τη. και θα έκανε τις αρμοδιότητες, που, θα διενεργούσε τις έρευνες που αφορούν τους υπηκόους τους. Σε ό,τι αφορά την ε, ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διαφόρων χωρών και αυτή οργανώθηκε μέσω διαφόρων συνεδριάσεων που είχαμε στα πλαίσια της Eurojust. Εγώ έκανα κάποιες ε, αναλύσεις για το συριακό πορτοφόλι, αυτόν τον τρόπο διακίνησης χρημάτων και ε, είδα ότι πολλοί Βέλγοι επίκοοι έστειλαν χρήματα από το Βέλγιο. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούμε το άρθρο 7 της ε, Σύμβασης του Σέγγεν της 29ης Μαΐου του 2000 Εκεί καταγγέλουμε αμέσω τα, τα πραγματικά περιστατικά στην αρμόδια δικαστική αρχή με το όνομα του αποστολέα. Επίση, στα πλαίσια τη καταπολέμη χρηματοδότηση των μεμονωμένων τρομοκρατών μαχητών, έχουμε διάφορα μέσα δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και θεωρώ ότι αυτά τα μέσα έχουν λειτουργήσει σχετικά εύκολα και καλά. Ένα άλλο παράδειγμα στη δικαστική συνεργασία στα πλαίσια χρηματοδότηση τη τρομοκρατία είναι η περίπτωση Lafarge τη γνωρίζετε. Βέβαια συνεχίζεται η έρευνα, η ανάκριση για το θέμα αυτό και παρόλο που είχαμε σημαντικές διαρροές στον τύπο για το θέμα αυτό δεν ε, μπορώ να σας δώσω πολλές πληροφορίες. Εγώ έχω αναλάβει το θέμα ε, το δικαστικό στο, στο Βέλγιο και πολλές φορές από τον τύπο μαθαίνουμε ε, μερικά στοιχεία της έρευνας που γίνεται είτε στη Γαλλία είτε εδώ στο Βέλγιο. Οπότε πολλές πληροφορίες έχουν ήδη διαρρεύσει. Η Όμιλος Λαφάρς είναι μια πολυεθνική εταιρεία τσιμέντο βιομηχανίας με εργοστάσιο στη Συρία που μάλιστα το είχε εγγενιάσει και είχε επενδύσει περίπου 700.000 ευρώ αλλά δυστυχώς ατύχησε η Λαφάρς γιατί το εργοστάσιο εγγενιάστηκε το 2010-2011 και λίγο αμέσως μετά ξεσπάσε ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία ο Όμιλος Λαφάρζ ε, είναι ύποπτος αυτή τη στιγμή για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων στη Συρία, πληρώνοντας κάποιους που μπλόκαραν, αυτούς, ε, ε, μπλόκαραν τους δρόμους πρόσβασης στη τσιμεντοβιομηχανία και ανταμείβοντας τις τρομοκρατικές οργανώσεις για να προστατεύσουν το αργοστάσιο τους σε ό,τι αφορά τις γαλλικές αρχές, τις δικαστικές αρχές, ε, έγινε καταγγελία από τους ε, ε, πρώην υπαλλήλου τη Λαφάρζ από τη Συρία κυρίω. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τι δικαστικέ αρχέ, γιατί τα πράγματα λίγο διαφορετικά για τι μυστικέ υπηρεσίε, να σα πω ότι είμαστε λίγο ενημερωμένοι για το τι συμβαίνει σε ό,τι αφορά την συρια ιρακινη ζώνη σε διάφορε περιπτώσει. Υπάρχουν διάφορε φήμε, αλλά συγκεκριμένα από τα στοιχεία για το τι συμβαίνει στο, στη Συρία και στο Ιράκ ε, δεν έχουμε πολλά στοιχεία σε ό,τι αφορά τη Λαφάζ. Να σας πω ότι το θέμα αυτό είναι ιστορικό της Γαλλίας γιατί ήταν γαλλική εταιρεία και Γάλλος ο διευθυντής με βάση το Παρίσι τότε και άρα δεν μας απασχόλησε ιδιαίτερα το θέμα αυτό αλλά να σας πω ότι βασικός μέτοχος, ο μέτοχος αναφοράς της Λαφάζ ήταν η Λαουντίν Μπέλζ, η οποία είναι γνωστή γνωστή εταιρεία η οποία ζήτησε να γίνουν έρευνες ε, ζητήθηκε μάλλον να γίνουν έρευνες στη ΖΕΜΠΕΛ δεδομένου ότι και το Βέλγιο θα ήταν θα αντιφερόταν. Γιατί αν ελέγχθησε απόφαση από τους μετόχους να διατηρήσουν την δραστηριότητά τους ε, στην ε, Συρία, Ενδεχομένω τελικά αυτή η χρήση να οδηγούσε σε χρηματοδότηση οργανώσεων όπω και η ΔΕΣ. Τρία λεπτά. Τρία λεπτά έχω ακόμα. ναι. Άρα, τάχιστα αποφασίσταμε να γίνει κοινή ε, έρευνα με τις γαλλικές αρχές για το θέμα αυτό. Και το σύστημα αυτό των, κοινων, των κοινών ερευνών ήταν πάρα πολύ πρακτικό ό,τι αφορά τη συνεργασία των δικαστικών αρχών, γιατί το, η γαλλική έρευνα συμπλήρωνε την βαλγική και έτσι ένα τμήμα των πορισμάτων της γαλλικής έρευνας θα χρησιμοποιηθούν και για τη βελγική ε, δικαστική αγωγή. Άρα λοιπόν αυτό αποτελεί ένα παράδειγμα τη επικοδομητική συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Και να σα πω ότι στην Βελγική Εισαγγελία λάβαμε πολλέ αποφάσει από ευρωπαϊκέ έρευνε, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία και σε γενικέ ε, γραμμέ πρέπει να σα πω ότι είναι εύκολη η εκτέλεση των αποφάσεων αυτών και γρήγορη. Δεν έχουμε ιδιαίτερε δυσκολίε δυσκολίες ό,τι αφορά την εκκλησιμότητα και τη συνεργασία τη δικαστική σε ευρωπαϊκό επίπεδο εντάχει τώρα σε ό,τι αφορά την προσέγγιση μέσω της χρηματοδότησης έχει νόημα. Έχουμε κάποιον ο οποίος είναι ύποπτος, για παραδείγμα, για μετάβαση στα σύνορα μεταξύ Συρίας και Ιράκ. Γίνεται λοιπόν μια οικονομική ανάλυση σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο άτομο και τον περίγυρο του. Και αυτό μου δίνει τη δυνατότητα να καθορίσω κατά πόσον έχει πάρει χρήματα κάπου στα σύνορα μεταξύ Συρίας και, Τουρκίας και χρησιμοποιείται λοιπόν το στοιχείο αυτό σε ό,τι αφορά την αναχώρηση του από τη Συρία και η μέθοδος των αλλαδαπών μαχητών του FTF και της οικογένειας του υπόπτου. αν για παράδειγμα δεν έχω νέα του για δύο έτη. Διαπιστώνουμε για παράδειγμα και υποθέτουμε ότι ενδεχομένω ε, να είναι σημαντική αυτή η πληροφορία σε περίπτωση που κάποια στιγμή επιστρέψει στη βελγική επικράτεια και σε διάφορα θέματα τρομοκρατίας ε, μπορούμε να εξετάζουμε περιπτώσεις πλαστών εγγράφων, γιατί υπάρχει περίπτωση πόρων που μεταφέρονται χωρίς λόγο σε διάφορες χώρες. Ελβετία, Γαλλία, Αγγλία, οι οικονομικές αυτές έρευνες μας δίνουν την δυνατότητα να διαπιστώσουμε ότι πρόκειται για πλαστά έγγραφα. Να σας πω για δύο λεπτά για τα νομοθετικά εργαλεία, πολύ χρήσιμα, αλλά όχι σε ό,τι αφορά την πρόληψη των ε, τρομοκρατικών χτυπημάτων και επιθέσεων, γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει κανένας σύνδεσμος χρηματοδότησης μεταξύ της μονάδας που θα διαπράξει την επίθεση και της ε, που έχει οργανώσει το χτύπημα σε επίπεδο δικαστικής ε, συνεργασίας. Να πω το εξής, είναι ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί σχετικά καλά Σίγουρα πολλά ακόμα θα πρέπει να βελτιωθούν, πολλά στοιχεία ακόμα θα πρέπει να βελτιωθούν, αλλά να σας πω ότι είμαι σχετικά ικανοποιημένο στην παρούσα από αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέγει η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαγιανίνη για την παρουσίαση αυτή. Πάρα πολύ πυκνή και αυτή. Και πάρα πολλά συγκεκριμένα παραδείγματα μας δώσατε, συγκεκριμένα περιστατικά δικαστικές αποφάσεις ε, ή περιπτώσεις όπου χρειάστηκε η κρίση σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ε, δηλώσεις αυτές που κάνατε για τον ε, μηχανισμό δικαστικής συνεργασίας ο οποίος λειτουργεί καλά από ό,τι μας είπατε και το θέμα της διάστασης μάλλον της χρηματοδότησης των αλλοδαπών μαχητών και την απόδειξη Ζωή μετά από πολλά χρόνια σε ορισμένε περιπτώσει και να δώσω το λόγο πάρα αυτά στην κυρία Γκόμε, η οποία είναι συντονίστρια των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Αγαπητοί συνάδελφοι σας, παρακαλώ να είστε σύντομοι στι ερωτήσει σα, γιατί ο κύριο Μαλανίνη θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στα επόμενα 10 λεπτά. Κύριε Μαλανίνη, η κυρία Γκόμε, όταν μιλάτε για διακίνηση για τη Western Union και το καθεξής. Είχατε συνεργασία και για την Αουάλα. Είχατε ε, ευκαιρία συνεργασίας ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα άτομα και τι μπορείτε να μας πείτε για το σύνδεσμο και τη σύνδεση με τα κυκλώματα εγκλήματος, οργανωμένου εγκλήματος που συνδέονται σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότησή τους και με τα τρομοκρατικά κυκλώματα σε ό,τι αφορά κυρίως ε, το λαθρεμπόριο ε, ναρκωτικών, όπλων και ανθρώπων. Και τέλος, να σας πω σε επίπεδο προσελτισμού, σε επίπεδο του Βελγίου. Προσελτισμό για άδειε προφανώς πράξεις. Νομίζω ότι το Βέλγιο έχει λάβει κάποια συγκεκριμένα μέτρα. Τι μπορείτε να μας πείτε από πλευρά των δικαστικών φορέων. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά την πρώτη σας ερώτηση. Η σχέση μεταξύ τρομοκρατίας στο Βέλγιο και της, του οργανωμένου εγκλήματος. Έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει τέτοια σύνδεση, τέτοια σχέση. Να σας εξηγήσω. Θεωρώ ότι η μοναδική σχέση που υπάρχει μεταξύ των ε, τρομοκρατών, τους οποίους βλέπω συχνά, και του οργανωμένου εγκλήματος, των κοινών εγκληματίων, είναι ότι συχνά ξεκινάνε από μικρά παραπτώματα. Έχουν δικαστικό παρελθόν, έχουν συχνά ένα μητρό. Άρα είναι γνωστή στη δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά τα πλαστά έγγραφα. Έχουμε διαπιστώσει ότι οι τρομοκράτες ε, χρησιμοποιούν ε, τα συνηθισμένα κυκλώματα για την ε, κατασκευή και την ε, παρανομή, την παραχάραξη γράφων. Τα κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος φαίνεται ότι είναι προφανή. Αλλά οι τρομοκράτες έχουν σύνδεση. Μάλλον συχνά οι τρομοκράτες έχουν περάσει και από κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος και έχουν τις ε, επαφές τους και εκεί. Αυτό που σημαίνει όταν κάποιος ε, διαπιστώνουν ότι είναι τρομοκράτης στους κόλπους των, του οργανωμένου κλίματος είναι να απομακρυνθούν από αυτό συχνά, γιατί φοβούνται ότι θα κατηγορηθούν και αυτοί. Σε ό,τι αφορά την τη χρηματοδότηση του θρησκευτικού προσελτισμού, την οποία αναφέρατε, ο προσελτισμός δεν αποτελεί έγκλημα. Άρα η διανομή και διάχυση κάποιων ιδεών δεν αποτελεί παράπτωμα και αδίκημα. Στο Βέλγιο παρακολουθούμε συχνά τις ε, εταιρείες μικροδοσκοπικού χαρακτήρα της ASBL ε, σε ό,τι αφορά τον προσελκτισμό που ασκούν. Και όταν υπάρχουν δωρεέ, υπάρχει ανησυχία σε πολλέ περιπτώσει ότι θα διοικητευτούν στη χρηματοδότηση παρανόμων δραστηριοτήτων. Υπάρχει λοιπόν συνεργασία μεταξύ των αρχών, των ε, οργανώσεων με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και η παρατηρήση και η υποπτή αυτή γίνεται και από τα αρμόδια Υπουργεία για τις Κοινωνικές Υποθέσεις γίνεται έλεγχο ε, των λογαριασμών, κατά σωστοί λογαριασμοί, τηρούνται σωστοί λογαριασμοί, ε, κοιτάμε πού διοχετεύονται τα χρήματα αυτά. Αλλά φυσικά τα χρήματα που περνάνε από χέρι σε χέρι ε, στο τζαμί. Αυτά φυσικά οι δικαστικές αρχές δεν μπορούν να τα έχουν υπόψη τους. Εδώ βασιζόμαστε πολύ στις ε, μεσικές υπηρεσίες για να μας ε, ενημερώνουν το τι συμβαίνει στα μέρη αυτά όπου δεν έχουμε πρόσβαση εμείς ως δικαστικές αρχές. Η Western ε, Union συνεργάζεται. Αυτό το επιβεβαιώνω. Κάθε φορά που είχαμε έτοιμα για έρευνα στην Western Union, πρέπει να σας πω ότι η ερώτηση ήταν άμεση. Αν δεν, είμαι, αν δεν κάνω λάθος, είναι θηγατρική Αμερικανική εταιρεία και υπάγεται σε Αμερικανικό δίκαιο σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία. Είναι πολύ καλή η συνεργασία. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και να δώσω το λόγο στην Ελγα Στίβεν, η οποία είναι μία από τις δύο συνεισηγητρίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι ω ε, συνεισηγητρία καθήκον μου να προτείνω κάποια συγκεκριμένα μέτρα με μια προστιθέμενη αξία. Καταρχά, πιστεύετε ότι υπάρχει σχέση μεταξύ τη ε, μαύρη αγορά και τη τρομοκρατία και υπάρχει μήπω μια ροή χρημάτων που την ξεχνάμε, υπάρχει κάποιο σύνδεσμο που το ξεχνάμε και πώ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις ε, τρομοκρατικές οργανώσεις που χρηματοδοτούνται μέσω της μαύρης αγοράς. Ε, σε ό,τι αφορά επίσης το, κρυπτα, το συνάλλαγμα, τα κρυπτονομίσματα, ε, τι γίνεται με αυτά σε ό,τι αφορά και πάλι τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Σας ευχαριστώ πολύ lien entre le marché noir et plus particulièrement... Μεταξύ euh, μαύρης αγοράς ε, και και αγορά ε, εργοτέχνη υπάρχει τέτοιο σύνδεσμο ε, πολιτισμική, αν θέλετε Ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή η σύνδεση με τη τρομοκρατία. Είχα κάνει μια έρευνα στην Ισπανία όπου υπήρξε μια σχέση ε, μεταξύ έργων τέχνης και τρομοκρατίας. Μας είχαν απαντήσει λοιπόν πάρα πολύ γρήγορα στο έτοιμά μας για πληροφορίες. Σε επίπεδο Βελγίου ξέρω ότι υπάρχει αυτή η σύνδεση, αλλά εγώ σε ένα γραφείο κάθομαι, έναν υπολογιστή έχω. Έχουμε θέσει προφανώ διάφορε ερωτήσει σε διάφορε υπηρεσίε, αλλά σε επίπεδο Βελγίου δεν έχουμε διαπιστώσει να υπάρχει τέτοια σύνδεση. Υπάρχει όμως ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο το θέμα αυτό και το έχουμε θέσει λοιπόν σε επίπεδο Ισπανία. Σε ό,τι αφορά το κρυπτονομίσματα, είναι η επόμενη πρόκληση αυτή για τη χρηματοδότηση τη ε, τρομοκρατία και του οργανωμένου κλίματο. Σα ε, ομολογώ ότι στην παρούσα φάση δεν ξέρω πώ θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό. Είναι πάρα πολύ πολύ σύνθετο και εδώ πάλι υπάρχει αυτή η εξωτερική διάσταση. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα πρέπει να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε και τι δεν θέλουμε να κάνουμε σε ό,τι αφορά την πρόσβαση ε, σε βάση δεδομένων όταν είναι κανεί στο εξωτερικό. Μίλησε και ο κ. Μπριζά για το θέμα αυτό και θα ήθελα να σας πω, αν μου επιτρέπετε, πέρα από το πλαίσιο τη συζήτησή μα σήμερα, ότι αν υπάρξει, αν υπάρχει κάτι στο οποίο θα πρέπει να εργαστούμε για να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία γενικά είναι η πρόσβαση των δικαστικών αρχών της Ευρώπης σε στοιχεία και δεδομένα τρίτων χωρών. Και κυρίως αναφέρομαι και από την άλλη πλευρά των Αντικατοικού, στις, ε, μάλλον αναφέρομαι σε αυτό που ισχύει στη ΣΥΠΑ. Εκεί υπάρχει τέτοια πρόσβαση. Γιατί εξαρτώμαστε από την καλή θέληση των Αμερικανικών αρχών σχεδόν τώρα μας ε, Είχαμε έναν ύποπτο για βίες ε, ενέργειες. Ή, είπα, χωρίς να τους ζητήσω καν, μου έστειλαν όλο το φάκελο του facebook του ατόμου αυτού Εγώ προφανώς και χαρικά ιδιαίτερος και είπα ζήτω, αλλά να σας πω την αλήθεια, ότι στην περίπτωση που ένα δικαστή θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να λάβει τα στοιχεία αυτά, σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενδεχομένω να μην τα είχαμε πάρει τα στοιχεία. Είναι πολύ δύσκολα όλα αυτά και πολύ σύνθετα. Αλλά ε, αν ε, ω αρχέ δίωξη χρειαζόμαστε τα στοιχεία αυτά, υπάρχει το θέμα τη πρόσβαση στα δεδομένα. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεαλισμό αλλά και για τις διευκρινήσεις και για τις απαντήσεις βεβαίως στις ερωτήσεις των συναδέλφων. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαλανίνη με την εξαιρετική του παρουσίαση σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή δεδομένων δεν είναι κάτι που αμφισβητεί κανείς, ούτε οι συνσυνηγήτριε ούτε τα μέλη της Επιτροπής αυτής. Είναι ένα ζήτημα που βρίσκεται πραγματικά στο πυρήνα της Επιτροπής μας. Δεν το θίξατε, αλλά σε σχέση με τις με την δικαιοδοσία των διαφόρων υπηρεσιών. Μπορέσαμε να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις. Θίξαμε το ζήτημα της αγαστής συνεργασίας. Έχετε υπόψη σας κατά πόσο πρόκειται για μια προτεραιότητα για τα κράτη-μέλη η καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι ένα από τα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ σε κάθε περίπτωση όμως τον κύριο Μαλανινή για την συνεργασία του. Συμφωνούμε ότι εργαζόμαστε σε μια πρόταση νέων κανονισμών Αποκινούμε τον κύριο Μαλανινή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Mes chers collègues, Προτείνω να περάσουμε τώρα στο τρίτο σημείο της σημερινής μας ημερήσιας διάταξης. Να καλωσορίσουμε με μεγάλη χαρά τον Επίτροπο Πια Μοσκοβίση. Θα μας μιλήσει για τις ε, διαφορετικές προτάσεις που άπτονται των εργασιών της δικής μας Επιτροπής ενάντια στην χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ένα ζήτημα το οποίο μας παρουσίασε μόλις προηγουμένως ο κ. Μαλανίνη, κάτι που αφορά μόνο το Βέλιο αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη. Υπάρχουν εργαλεία που λειτουργούν και εδώ μαζί με τον Πιέρ Μοσκοβισή θα μιλήσουμε για τον έλεγχο των χρημάτων των μετρητών του ρευστού στην Ευρώπη για την χρήση της απάτης καρουζέλ, της απάτης του ΦΠΑ στην υπηρεσία της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία και θα είναι βεβαίως οπωσδήποτε χρήσιμο αγαπητέ Πιέρ αν καταφέρετε να μας παρουσιάσετε λίγο πόσο ανασχηματισμός των κανονισμών θα μας βοηθήσει να καταπολεμήσουμε αυτήν την απάτη σχετικά με το ΦΠΑ. Η παρουσίαση του ανασχηματισμού αυτού για τους κανονισμούς που αφορούν στην απάτη του ΦΠΑ είναι η πιο μαζική. Μιλάμε για 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι μία από τις αρχαιότερες μεθόδους απάτης και ο ανασχηματισμός των κανονισμών στα πλαίσια της Επιτροπής που προτείνεται θα τεθεί σε εφαρμογή το 2020. Έχετε ζητήσει από τα κράτη αλλά και από την δική μας Επιτροπή να σας συμπαρασταθεί. Έχουμε πλήρη συνείδηση ότι η κοινή μάχη ενάντια στην τρομοκρατία άπτεται της αρμοδιότητας πολλών επιτρόπων και αν θέλουμε πραγματικά να πατάξουμε την ε, πληγή αυτή που έχει βλάψει ιδιαίτερα τη δική μας χώρα, τη δική μου και τη δική σας, ε, τη Γαλλία, είναι ανάγκη να εντείνουμε την ε, συνεργασία μας. Αγαπητέ Επιτρόπε, λοιπόν, σας προτείνω να πάρετε το λόγο για 15-20 λεπτά και αν είστε σύμφωνος να απαντήσετε με τη λεγόμενη μέθοδο ping-pong, ε, δηλαδή κάποιος θα σας κάνει μια ερώτηση και εσείς θα απαντάτε άμεσα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητή Ναταλή Γκρισμπέκ, ε, κυρίες και κύριοι αντιπρόεδροι, κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτέ. Δεν είμαι α, ο καταρχήν αρμόδιος επίτροπος για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αλλά στο δικό μου χαρτοφυλάκιο έχω πολλές αρμοδιότητες που είναι συναφείς ε, εισιδέονται κατά κάποιο τρόπο με το θέμα της χρηματοδότησης τρομοκρατίας Γι' αυτό και δεχτήκα ευχαρίστω στην πρόσκλησή σας και είμαι έτοιμος να απαντήσω στις απορίες στα μέτρα των αρμοδιοτήτων μου βέβαια. Εν είδη εισαγωγής, θα ήθελα να ξεκινήσω με μια ε, περίπτωση ανεκδοτικά, δεν είναι καθόλου αστείο βέβαια. Πριν από λίγες μέρες ένας πελοπόλης αντικέρ, Ισπανός, συνελήφθη στη Βαρκελόνη για την υποτιθέμενη συμμετοχή του σε ένα τεράστιο λαθρεμπόριο προϊόντων αρχαιοκαυπηλείας Και μάλιστα η έρευνα έδειξε ότι πολλά έργα τέχνης ε, που είχαν ε, κλαπεί και λετηθεί από ε, λιβικούς αρχαιολογικούς χώρους από την οργάνωση, τη γνωστή τρομοκρατική οργάνωση ΝΤΑΕΣ, η Ισλαμικό κράτος και το λαθρεμπόριο αυτό αρχαιολογικών αντικειμένων και αρχαιοτήτων στόχο είχε τη χρηματοδότηση της Ισλαμιστικής τρομοκρατίας. Και μάλιστα αυτή η υπόθεση μας δείχνει πόσο σημαντικός είναι ο ο αγώνας μας για να εξαντλήσουμε, να στεγνώσουμε τους οικονομικούς πόρους των τρομοκρατών, ώστε να μην μπορούν να χρηματοδοτήσουν ε, μεγάλου ελληνικού τρομοκρατικέ επιθέσει. Οι πόροι τη ε, τρομοκρατία είναι πολύ άριθμοι. Είναι καταρχήν το εμβόλιο προϊόντων αρχαιοκαπηλεία, ε, ελευθερεμπόριο ναρκωτικών, οργανωμένο έγκλημα και μερικέ φορέ είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο θέματα. Επίση έχουμε τη φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή και υπάρχουν και εκεί κάποιες διακλαδώσει και συνάφειες με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Οπότε έχουμε πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες για τη χρηματοδότηση των τρομοκρατών. Αναχαιτίζοντας αυτές τις δυνατότητες θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε τα σχέδιά τους και να παρεμποδίσουμε τις βαναυσότητες που διαπράττουν μερικές φορές στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και μάλιστα πολύ πρόσφατα βυθιστήκαμε στο πέθος από τέτοιο έγκλημα. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ιδιαίτερα προσιλωμένη στο θέμα αυτό και μάλιστα ήδη το Φεβρουάριο του 2016 με ε, πρόταση των γαλλικών αρχών υπέβαλα ένα σχέδιο δράσης προκειμένου να ενισχυθεί ο αγώνας μας κατά τη χρηματοδότηση τρομοκρατία. Και ένα πυλώνα αυτού του σχέδιου δράση ήταν ακριβώ να μειώσουμε τι πηγέ εσόδων των τρομοκρατικών οργανώσεων. Και στο πλαίσιο αυτό, ω Επίτροπο Αρμόδιο για τα Τελωνία και τη Φορολογία, Υπέβαλα πρόσφατα προτάσει προκειμένου να ενισχύσουμε του τελωνιακού ελέγχου σε στρατηγικού τομεί. Θα σας του αναφέρω όσον νούπο. Και επίσης ε, να ευθύσουμε μέτρα για να καταπολεμήσουμε καλύτερα την φοροδιαφυγή. Και σε αυτό το θέμα θα αναφερθώ σε λίγο. Ε, στα θέματα των τελωνιακών ελέγχων ε, έχουμε υποβάλει στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύο προτάσει. Μία για τον έλεγχο των πολιτιστικών αγαθών, ώστε να προ να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση του προϊόντος, το, της διακίνησης προϊόντων αρχαιοκαπηλείας στην ευρωπαϊκή αγορά και ε, προϊόντων πολιτιστικής κληρονομιάς ε, που χρηματοδοτούν την τρομοκρατία και η δεύτερη πρόταση αφορά τον έλεγχο των μετρητών ή ρευστών που μπαίνουν και βγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, καταρχήν, στον έλεγχο τη διακίνηση αρχαιοτήτων ή αρχαιολογικών αγαθών, όλοι συγκλονιστήκαμε από την καταστροφή και τη λελασία αρχαιολογικών χώρων ανεκτήμητης αξίας από το Ισλαμικό κράτος και μάλιστα ήταν συμβολική σημασία σε αυτή η αρχαιολογική χώρη που καταστράφηκαν. Επίσης είναι εξίσου συγκλονιστικό ότι κάποια τέτοια αγαθά πολιτιστικά, αρχαιολογικά διακινήθηκαν παράνομα για να χρηματοδοτήσουν τρομοκρατικές δραστηριότητες. μάλιστα στις 30 Μαρτίου το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών εξάρθρωσε ένα διεθνές κύκλωμα διακίνησης ε, αρχαιοτήτων που προορίζονται για επαναπόληση στην ευρωπαϊκή αγορά. Πρόκειται για ψηφιδωτά, Σαρκοφάγου, αγγεία που είχαν ληλετηθεί από το Ισλαμικό κράτος στη Λιβύη. Και μάλιστα και εγώ προσωπικά ήμουν μάρτυρας ε, πριν από ένα χρόνο μιας κατάσχεσης από, από τα γαλλικά τελωνία στο αεροδρόμιο του Ρουασί πολιτιστικών αγαθών που ληλατήθηκαν και που κατά πάσα πιθανότητα προέρχονταν από την περιοχή της Ιρακ Παλαιστίνο-Συριακής σύγκρουσης. Γνωρίζουμε την πρόκληση που αποτελεί αυτό το λαθρεμπόριο αρχαιοτήτων και αρχαιολογικών προϊόντων. Και δεν είναι μόνο το θέμα τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία, γιατί δεν απευθύνονται και δεν προορίζονται μόνο σε αυτή ε, τέτοια διακίνηση προϊόντων αρχαιοκοπηλία ε, χρηματοδοτεί και το οργανωμένο έγκλημα ή χρησιμοποιείται για νομοποίηση εσόδων από παράνομε δραστηριότητε. Είναι απαράδεκτο τέτοια προϊόντα πολιτιστικά που έχουν εξαχθεί παράνομα από τη χώρα προέλευσης να εισέρχονται και να κυκλοφορούν ελεύθερα, ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι από τι σημαντικέ δεσμεύσει που αναλάβαμε να προστατεύσουμε ε, και σε διεθνέ επίπεδο την αρχαιολογική, παγκόσμια αρχαιολογική κληρονομιά και μάλιστα όπω αυτή προσδιορίζεται στην UNESCO και με βάση τα κριτήρια αυτή τη οργάνωση. Και, και αυτό τον Ιούλιο του 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτησε μια πρόταση κανονισμού που επιβάλλει τελωνιακού ελέγχου στην εισαγωγή των κυρίω πιο ευαίσθητων πολιτιστικών αγαθών. Για ένα ε, σημαντικό ρυθμό αυτών των έργων ε, αρχαιολογικών ή ε, άνω των 150 ετών. Μιλούμε για χειρόγραφα, για παλιά βιβλία ή για ε, αντικείμενα που προέρχονται από το διαμελισμό των κάποιων μνημείων. Οι εισαγωγείς θα πρέπει να αποδείξουν τον, ε, την νόμιμη προέλευση των προϊόντων που διαθέτουν. Αυτή η θέση είναι το αποτέλεσμα μιας παγκόσμιας συνειδητοποίησης του κινδύνου που συνιστά αυτό το λαθρεμπόριο έργων τέχνης και έχουμε πολλαπλές εκκλήσεις από διεθνείς οργανώσεις, από κράτη-μέλη και από άλλες συνελεύσεις μετά την καταστροφή αρχαιολογικών χώρων και μνημείων που διαπράχθη από τον ΤΑΕΣ, από το Ισλαμικό κράτος. Και αυτή η πρόταση αυτή τη στιγμή συζητάται στο Συμβούλιο και στις κοινοβουλευτικές επιτροπές Διεθνούς Εμπορίου και Προστασίας των Καταναλωτών. Και μάλιστα προσβλέπω στη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευελπιστώ ότι το, οι εργασίες θα διεκπαιρεωθούν πριν τι ευρωεκλογέ του 2019. Θέλω να επισπεύσουμε τι εργασίες ώστε να υιοθετηθεί αυτή η πρόταση το συντομότερο δυνατό. Γιατί ε, το να περιμένουμε μέχρι τον Ιούνιο, Ιούλιο 2019 είναι μεγάλο διάστημα για ένα τέτοιο κείμενο που ούτως ή άλλως ε, μας βρίσκει σύμφωνο, σύμφωνος ως προς την ουσία. Καλό θα ήταν λοιπόν να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Απέναντι στην όλο και μεγαλύτερη ευρηματικότητα των εγκληματικών και τρομοκρατικών κυκλωμάτων θα πρέπει να επικαιροποιήσουμε τους και να ενισχύσουμε τους κανόνες για την είσοδο και έξοδο ρευστών στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι το αντικείμενο τη δεύτερη πρόταση που θα σα παρουσιάσω γιατί οι τρομοκρατικές και εγκληματικές οργανώσεις έχουν βρει τρόπους να παρακάμψουν τους ισχύοντες κανόνες που διέπουν τον έλεγχο των κινήσεων ρευστού χρήματος, είτε στέλνοντας ταχυδρομικά ε, μετρητά, είτε χρησιμοποιώντας ε, το χρυσό ή τις προπληρωμένες κάρτες ε, που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και έχουν αξίσει ουσιαστικά ρευστού χρήματο. Για παράδειγμα, το 2015 τα γαλλικά τελωνία εντόπισαν αδήλωτα μετρητά στο αεροδρόμιο Ρουασί, καθώς και ε, χρυσό από ταχυδρομικές και εμπορευματικές αποστολές ύψους ε, άνω των 9,2 εκατομμυρίων ευρώ. Οπότε προτείναμε να τροποποιήσουμε τον ισχύοντα κανονισμό ενισχύοντας τους ελέγχους που ισχύουν για ποσά άνω των 10.000 ευρώ που στέλνονται ε, μέσω ε, ταχυδρομείου. Διευρύνουμε τον ορισμό του ρευστού των μετρητών ώστε να περιλάβουμε και τις προπληρωμένες κάρτες και το χρυσό και δημιουργούμε έναν πιο απλό και στιβαρό μηχανισμό για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ε, αρχών ε, μυστικών υπηρεσιών και τελωνιακών εθνικών αρχών και των ε, εθνικών τμήματων οικονομικών υπηρεσιών. Επίσης, επιτρέπουμε στις αρμόδιες αρχές για ποσά κάτω των 10.000 ευρώ να γίνεται τέτοιο έλεγχο, εφόσον υπάρχουν εύλογε υποψίε ότι πρόκειται για τρομοκρατική δραστηριότητα. Έτσι αυξάνουμε τη δυνατότητα εντοπισμού από τι αρμόδιε Εθνικέ αρχέ τρομοκρατικών ή ε, εγκληματικών κυκλωμάτων που δημιουργούν, χρησιμοποιούν μεγάλε ε, ε, χρημάτων για να περάσουν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή ε, βρισκόμαστε σε φάση τριμερούς διαλόγου στην κοινοβουλευτική, ε, στις κοινοβουλευτικές επιτροπές ΕΚΟΝ και ΛΥΜΠΕ και ε, ελπίζω να καταλήξουμε στη συμφωνία μέχρι το καλοκαίρι. Επίση, προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη δυνατότητα, τις δυνατότητες και τις ικανότητες των τελωνιακών αρχών να εντοπίζουν τους κινδύνους και ετοιμάζουμε μια ρηξικέλευθη μεταρρυθμίση του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου των εισαγωγών προκειμένου να ενισχύσουμε την ασφάλεια των εμπορευμάτων, να εντοπίσουμε τις παράνομες διακινήσεις, εντοπισμό εκρηκτικών, ναρκωτικών, όπλων και διάφορα είδη λαθρεμπορεί, όπως είναι ε, τσιγάρα και προϊόντα παραποιημένα, μαϊμούδες. Η μεταρρύθμιση του συστήματο ελέγχου εισαγωγών και τα νέα μέτρα του Τελωνιακού Κώδικα θα έχουν κέρια σημασία για να αντιμετωπίσουμε τις, τους διασυνοριακούς κινδύνους ε, και τους κινδύνους στα εξωτερικά σύνορα. Επίση, είναι σημαντική η στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την κατά την προετοιμασία του επόμενου πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου. Γιατί όλα αυτά προϋποθέτουν ε, πόρους και χρηματοδότηση των τελωνίων. Είναι φιλόδοξη αποστολή της και θα πρέπει, χάρη στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, να προβλεφθούν τα απαραίτητα μέσα ε, και όχι απλώς συμβαλωματικά για να ανταπεξέλθουν στο έργο τους. Σε ό,τι αφορά την, ε, το παράνομο εμπόριο έργων τέχνης και τις παράνομες μεταφορές κονδυλίων, το θέμα της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής επίσης είναι πολύ σημαντικό για τις τρομοκρατικές και εγκληματικές οργανώσεις. Και από την αρχή των, ε, του, της εντολής μου, ο έλεγχος της φοροδιαφυγής και το πώς θα κόψουμε, θα στεγνώσουμε τις πηγές εσόδων των τζιχαντιστών είναι σημαντικό ε, σημαντική προτεραιότητά μου και μάλιστα οι δικαιοδοσίες που δεν σέβονται τους διεθνείς κανόνες για την χρηστή ε, φορολογική διακυβέρνηση είναι σημαντικός και μάλιστα πολλές ε, χώρες του καταλόγου αυτού έχουν αναλάβει δέσμευση να σεβαστούν τις τι συστάσει μα και έχουμε πέραν τη μαύρη Λίστα και έναν γκρι κατάλογο αυτό το μεταβατικό χώρο που δήλωσαν ότι θα σεβαστούν του κανόνες. Θέλουμε ένα καλό επίπεδο παγκόσμια χρηστή φορολογική διακυβέρνηση για να αποφύγουμε καταχρηστική φορολογική διαφορά, συμπεριφορά μεγάλη κλίμακο. Επίση, να αποφύγουμε το ξέπλυμα τη βρώμικου χρήματος ε, και μάλιστα συγκεντρω... συνεργάζομαι με την αρμόδια επίτροπο για την καταπολέμηση τέτοιων, θεμα... τέτοιων συμπεριφορών. Αλλά δεν χρειάζεται να πάμε μόνο στο θέμα των φορολογικών παραδείσων για να διαπιστώσουμε φορολογική... φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή. Έχουμε αποδείξεις ότι οι τρομοκρατικέ και εγκληματικέ οργανώσει χρηματοδοτούνται από τη φοροδιαφυγή ακόμη και εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα έμεινα άναυδος ε, παρακολουθώντας δύο ε, ντοκιμαντέρ Δανών και Ολλανδών δημοσιογράφων πέρυσι τον Οκτώβριο που ε, παρουσίαζε τη χρηματοδότηση από ε, τζιχαντιστές ολόκληρων κλάδων ε, μέσω της ε, απάτης στο ΦΠΑ, διασυνοριακή απάτης, που ανέρχεται σε 50 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και θα ήθελα παρεμπιπτόντω να σας ε, συστήσω να παρακολουθήσετε αυτά τα δύο ντοκιμαντέρ που είναι πολύ κατατοπιστικά και μάλιστα είχαμε οργανώσει και ένα σεμινάριο με τους δημοσιογράφους που ε, δημιούργησαν αυτό το, το ντοκιμαντέρ και ήταν πολύ ενημερωτική η παρουσίαση. Επίση, τον περασμένο Οκτώβριο πρότεινα μια εκπάθρο αναδιατύπωση του συστήματο ΦΠΑ για να ανακόψουμε τέτοιε απάτε καρουσέλ. Με την πρόταση αυτή θα μειωθεί κατά 80% η και απάτη ΦΠΑ. Αυτή τη στιγμή το θέμα εξετάζεται στο Συμβούλιο και θέλει να δώσει στις, ε, στις εθνικές φορολογικές αρχές τα μέτρα για να καταπολεμήσουν τη διασυνοριακή απάτη στο ΦΠΑ και να ενισχύσει τη δυνατότητά τους για να καταπολεμήσει αυτό το θέμα της απάτης από το οργανωμένο έγκλημα. Οπότε θα πρέπει να συνεργαστούν οι εθνικές αρχές με την Όλαφ, τη Europol και την Ευρωπαϊκή Αγγελική Αρχή και νομίζω ότι ε, χάρη στις προτάσεις αυτές τα, τα κράτη-μέλη θα προσχωρήσουν σε αυτή την ιδέα της συνεργασίας γιατί η τρομοκρατία και η καταπολέμηση των ε, απατών στο ΦΠΑ είναι διασυνοριακά φαινόμενα. Χρειάζεται λοιπόν συνεργασία για να καταπολεμήσουμε την απάτη στο ΦΠΑ που χρηματοδοτεί τρομοκρατικά και εγκληματικά κυκλώματα. Για να ολοκληρώσω λοιπόν, η τρομοκρατία είναι ένα φαινόμενο που εξελίσσεται με τον χρόνο και αποκτά και πιο εξειδικευμένε μορφέ. Αρχαιολογικά αγαθά, ξέπλυμα χρήματο, φοροδιαφυγή, είναι πολλέ και διάφορε οι πηγέ χρηματοδότηση, οπότε και οι μηχανισμοί μα άμυνα θα πρέπει να προσαρμόζονται στι εξελισσόμενε προκλήσει. Βέβαια με τι προτάσει μα ε, ε, θα, θα καταφέρουμε ε, να μειώσουμε σε κάποιο βαθμό την τρομοκρατία μεγάλου κλίματος και θέλω να είμαι μετριόφρον βέβαια, αλλά με σταθερή και αμήλικτη φιλοδοξία θα προσπαθήσουμε να αναχαιτήσουμε αυτά τα θέματα της χρηματοδότησης. Βέβαια έχουμε πολύ έργο να κάνουμε ακόμη και θα ασχοληθείτε και εσείς με αυτό το θέμα της ριζοσπαστικοποίησης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται με αυτό το ζήτημα που έχει κέρει κεντρική σημασία και θα ήθελα να σας εκφράσω την απόλυτη διαθεσιμότητα μου και προθυμία μου και τη δική μου και των υπηρεσιών μου για να συνεργαστούμε στην πρόθεση αυτών των εργασιών σας ό,τι αφορά τις προτάσεις μου και επίσης είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε απορίες που σχετίζονται φυσικά με το χαρτοφυλάκιό μου και τις αρμοδιότητές μου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Επίτροπε. Αγαπητέ Πιέρ, για την πολύ συνοπτική αυτή και εκτενή παρουσίαση. Και για τα συγκεκριμένα παραδείγματα που μας δώσατε σε ό,τι αφορά τη σχέση μεταξύ οργανωμένου κλίματος, φοροαπάτης, απάτης ΒΠΑ και του τρομοκρατίας, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ήταν ε, σαφές ε, το μήνυμά σας, το ακούσαμε και στην ΙΜΚΟ και στην ΙΝΚΤΑ και σε άλλες ε, επιτροπές. Σχεδιάζουμε και συνάντηση με τον Επιτροπό για να μπορέσουμε να δαπανίσουμε τους πόρους εκεί που χρειάζονται, παρά το γεγονός ότι είναι περιορισμένοι αυτοί οι πόροι. Φυσικά κατά προτεραιότητα σε αυτά που απασχολούν τον Ευρωπαίο πολίτη σε μια σωστά οργανωμένη ασφάλεια. Και να δώσω το λόγο στους συναδέλφους για τις ερωτοαπαντήσεις. Να αναφέρω μόνο το εξή. Σε ό,τι αφορά αυτά που πετεκλίνονται, κύριε Επιτροπέ, για τις αρμοδιότητες. 40 χρόνια χρειάστηκαν για να καταλήξουμε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στη συνεργασία. Δυστυχώς μόνο συνεργασία. Αλλά Ποια είναι η άποψή σας για την διάφρυνση των αρμοδιοτήτων τη εισαγγελία, όχι μόνο για τέτοια χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Είναι λίγο α, ευρύ το θέμα, το ομολογώ αλλά συμμετέχετε στο σώμα των επιτρόπων. Παρά το γεγονό ότι ο καθένα έχει τι ε, κάθετε αρμοδιότητέ του, υπάρχουν και οριζόντια θέματα. Το λόγο έχει η κυρία Άννα Γκόμε, συντονίστρια τη Επιτροπή από του Σοσιαλιστέ για Δημοκράτε. Ευχαριστώ πολύ, Επιτροπέ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σα και νομίζω ότι πρωτού δαπανίσουμε τους πόρους θα πρέπει να τους βρούμε τους πόρους αυτούς. Κυρίως ό,τι αφορά πόρους που καταλήγουν σε εγκληματικές οργανώσεις και τρομοκρατικές οργανώσεις. Σε ό,τι αφορά το παράνομο εμπόριο, το λαθρεμπόριο ε, πολιτιστικών αγαθών. Σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, το Λουξεμβούργο, στην Ντουμπάι, Επισκεφθήκαμε το Λουξεμβούργο πρόσφατα και μας είπαν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από τους τελενιακούς ελέγχους. Σε ό,τι αφορά τα πολιτισμικά αγαθά, πώς γίνεται να αποθηκεύονται επί σειρά ετών. Το θέμα της ε, φοροαπάτης, ε, της απάτης σε καρουσέλ. Μιλάμε για δισεκατομμύρια, 50 δισεκατομμύρια είπατε. Και 10 δις απάτη από τους αμέσους φόρους κατανάλωσης. Η πρότασή σας ε, είναι στο τραπέζι του και ένα χρόνο και πλέον. Αυτή ήταν και ταινία, αυτό το ρεπορτάζ από τη Δανία και τη Ολλανδία ε, το διατίθεται από πέρσι τον Οκτώβριο. Και οι κυβερνήσει, οι οποίε βγαίνουν και λένε στου πολίτε ότι πολεμούν την τρομοκρατία δεν έχουν κάνει τίποτα. Αυτό πραγματικά μου φαίνεται περίεργο. Εγώ λοιπόν ρωτώ, ποια είναι τα κράτη-μέλη που μας μπλοκάρουν, που διστάζουν, που δεν αφήνουν να περάσουν τα μέτρα. Αγαπητή Άννα, λέει πρόεδρος, θα κοκκινήσει ο Επιτροπός. Κοιτάξτε, πρόεδρε, καταρχάς, να σας πω ότι και εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα είναι ανεξάρτητη υπηρεσία και θα έχει αρμοδιότητα να κάνει τέτοιες έρευνες για περιπτώσεις όπως είναι για παράδειγμα τι ιστοριακές απάτες. Και πάνω από τα 10 δισεκατομμύρια αυτά, προφανώ χρειάζονται διάφορε πρωτοβουλίε που έχουν ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι οποίε ε, όλε τον ίδιο σκοπό έχουν. Την ενίσχυση τη συνεργασία μεταξύ των ε, δικαστικών αρχών και την αναζήτηση νέων τρόπων καταπολέμησης της πιο σημαντικής απειλής σε ό,τι αφορά την παράνομη, τα παράνομα έσοδα. Η νέα εισαγγελία λοιπόν μπορεί να αποτελέσει μια πολύ σημαντική αρχή για την προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμα και από τις παρούσες αρμοδιότητες της. Επίσης η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να κοιτάξει και να καταπολεμήσει και τη θέμα της διαστημιακής τρομοκρατίας βάσει του άρθρου 126.4 και τα σοβαρά εγκλήματα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η τρομοκρατία και θα γίνει τον Σεπτέμβριο του 2018 θα δημοσιευτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία ανακοίνωση σε ό,τι αφορά τα μέτρα τα οποία προγραμματίζουμε να πάρουμε μέχρι το 2025 και κατά προτεραιότητα θα επικεντρωθούμε στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Εισηγγελίας και θα πρέπει φυσικά η ενεχόμενη διεύρυνση της εισαγγελίας να γίνει με συμφωνία όλων. Η ανακοίνωση λοιπόν το Σεπτέμβριο του 2018 μέχρι το 2025 σε ό,τι αφορά τα free zones ε, στους λεμμένες κτλ. Υπάρχει και ο Λαφσόλτς, ο οποίος είναι δήμαρχος και ήταν δήμαρχος και ε, με υπουργό οικονομικών Γερμανία. Οι υπηρεσίε μου λοιπόν έστειλαν ε, ρευματολόγια σε κάποια κράτη-μέλη για περιπτώσεις ε, ενδεχόμενης απάτης. Και υπηρεσίες όπως η Όλαφ, η Eurojust προσπαθούν και αυτές να αξιολογήσουν άλλα εγκλήματα. περιπτώσει παραχάραξη ή ξεπλήματο χρήματο. Όταν αυτά τα ερωτηματολόγια θα έχουν ε, απαντηθεί και θα έχουμε συλλέξει όλους τι απαραίτητε απαντήσει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει τι είδου επιπλέον ενεργείε χρειάζονται. Και επίσης θα συμμετάσχει ένεργα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τον ΩΣΑ και τα μέλη του για την κατάρτιση κατά των τριών γραμμών, καταρχάς για τις χώρες σε ό,τι αφορά τα free zones, για την καταπολέμηση των, ε, του παρανομού εμπορίου και για έναν ε, κώδικα δεοντολογίας, αν θέλετε. Και τα έγγραφα λοιπόν αυτά. Τα υπολογίζουμε, μάλλον τα λάβαμε το Σεπτέμβριο 2017. Ελπίζουμε να εγκριθούν σύντομα. Και θα τα εξετάσουμε στη συνέχεια και σε επίπεδο G20 ενδεχομένω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις απαντήσεις και να δώσω το λόγο στις δύο συνεισηγητρίες, την κυρία Μόνικα Χολμάιερ και την Έλγα ε, Στίβεν, συνεισηγητρία η Μόνικα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ σήμερα. Δεν ε, θα σας διευκολύνω με τις ερωτήσεις μου σε σχέση και με την, με την κυρία Γκόμες, γιατί στην Επιτροπή ΛΥΠΕ ασχολούμαστε πάρα πολύ συχνά με θέματα φοροαπάτης, απάτης ΦΠΑ και με άλλου είδους ε, απάτες σε ό,τι αφορά το τριμοποίηση εσόδων από παράνομες πηγές. Δυστυχώς δεν τα καταπολεμεί αυτά επαρκώς η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να σας αναφέρω δύο στοιχεία. Η Europol μας είπε ότι πέντε της χιλής των ε, παράνομα διακινούμενων πόρων ε, καταφέρει να εντοπίσει. Είμαστε πάρα πολύ απογοητευμένοι. Αν δηλαδή μόνο ένα πέντε της χιλίες καταφέρουμε να κατέσχουμε, ουσιαστικά έχουμε ξέφραγμα μπέλη. Αν οι εγκληματίες δρούν συντονισμένα. Κατά δεύτερον, έγινε μία ακρόαση εισαγγελέων για το θέμα ξεπλήματος χρήματος και ακούσαμε ότι 90% των εσόδων αυτών από παράνομες πηγές δεν φτάνει καν στα δικαστηρία και από αυτό το 10% 20 έως 30% τελικά καταφέρνει να καταδικαστεί. Πρόκειται για τάξεις μεγέθους που μας ανησυχούν ως βουλευτές. Γι' αυτό λοιπόν έχω τις εξής ερωτήσει να σε απευθύνω. Δεν έχουμε μόνο το εμπόριο πολιτισμικών αγαθών. Έχουμε και το πετρέλαιο, τα διαμάντια, το χρυσό και άλλα τέτοια υλικά τα οποία δυστυχώ εμπλέκονται σε πολλέ ε, παράνομε δραστηριότητε. Θα ήθελα να μα ενημερώσετε, αν γίνεται. Και κατά δεύτερον, υπάρχει εδώ και καιρό η ιδέα να δοθεί στην Ευρωπόλη η δυνατότητα να κάνει και ευρωπαϊκό FIU και να υπάρχει δυνατότητα με, να υπάρχουν άμεσε επαφέ με εθνικά τέτοια κέντρα. Τα εθνικά κέντρα συνεργάζονται μεν όλο και καλύτερα, αλλά η όλη ταχύτητα της συνεργασίας θα μπορούσε να ακολουθήσει το παράδειγμα της τρομοκρατίας των τελευταίων ετών, όπου τα πράγματα, πώς να το κάνουμε, επιτοχύνθηκαν. Γιατί η συνεργασία μεταξύ εθνικών FIU είναι πάντα χρονοβόρα και δύσκολη. Τρίτη ερώτηση. Στο πλαίσιο αυτό Ακούμε και πολλά ζητήματα για το e-evidence, τις τα ηλεκτρονικά αυτά τεκμήρια. Είτε πρόκειται για πληροφορίες υπηρεσιών ελέγχου, όπως και να έχει, για ύποπτες συναλλαγές, θα πρέπει να υπάρχει ταχύτερη ευρωπαϊκή ενημέρωση. Γιατί μόνο αν είναι καλή συνεργασία τελικά θα καταφέρουμε να πιάσουμε τα κυκλώματα, τα διασυνοριακά κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματο και χρηματοδότηση τη θερμοκρατία. Και κάπω αυτή η ταχύτητα μα απογοητεύει. Έχουμε και δαπανούμε τόσα πολλά χρήματα για να ελέγξουμε τι χρηματοοικονομικέ δραστηριότητε των πολιτών, των απλών πολιτών. Και εδώ που χάνονται δισεκατομμύρια σε παράνομε διαδικασίε, δεν κάναμε τίποτε. Ο Επίτροπος. Επίτροπε. Είναι αλήθεια ότι δεν απάντησα 100% στην κυριακό μές Η Επιτροπή παρουσίασε το 2016 μία πρόταση για να ενδυναμώσει τον εντοπισμό για τις απάτες σχετικές με το ΦΠΑ. Πρόκειται για νέες αρμοδιότητες και για νέες μεθόδους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με τη βοήθεια ψηφιακών μέσων. Γι' αυτό λοιπόν και η Κομισιόν προτείνει αυτήν την αυξημένη συνεργασία για την καταπολέμηση της απάτης από κοινού μαζί με τις υπηρεσίες ΟΛΑΦ και Europol κάτι το οποίο στηρίζουν στην πλειοψηφία τους και τα περισσότερα κράτη-μέλη. Το ερώτημα όμως ήταν διαφορετικό. Το ερώτημα της Γκομές είχε να κάνει με το ποιος εμποδίζει αυτήν την διασυνοριακή συνεργασία. Δεν μπορώ να ξεκινήσω εδώ μια λίστα. Η πρότασή μας όμως είναι πολύ συγκεκριμένη. Να αντιμετωπίζουμε το ΦΠΑ, να ορίζουμε το ΦΠΑ παντού με τον ίδιο τρόπο. Ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια διασυνοριακή αντιμετώπιση. Αν δεν υπάρχει μια κοινή αντιμετώπιση, έτσι προκύπτει αυτή η λεγόμενη απάτη καρουζέλ. Ιδού ο λόγος για τον οποίο εγώ προσωπικά δεν πιστεύω σε αυτούς τους μηχανισμούς γενικών χρεώσεων general charge κάποιες χώρες της κεντρικής Ευρώπης έχουν μια διαφορετική οπτική γωνία για πολιτικούς λόγους που πολλές φορές εμποδίζουν πρόοδο σε συγκεκριμένα σχέδια. Και εδώ και σε αυτό το σημείο η υποστήριξη του Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντική για την Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά εμένα, μπορώ να σας πω ότι είναι πολύ σημαντική η στήριξη του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Αυτό το σημείο λοιπόν είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και για τις δικές μου αρμοδιότητες. Πρόκειται για α, συγκεκριμένα μέτρα με συγκεκριμένα όρια σε ό,τι αφορά τις φυσικές α, α, χρηματικές ανταλλαγές αλλά και ανταλλαγές στο διαδίκτυο. Το 2008 προτείνουμε μια νέα στρατηγική για να μπορούμε να έχουμε πιο συγκεντρωμένο έλεγχο και να καλυτερεύσουμε την συνεργασία μεταξύ των διαφορών οικονομικών υπηρεσιών αλλά και της αστυνομίας. Τον Απρίλιο προτείναμε ένα πακέτο μέτρων για να καλυτερεύσουμε την αποτελεσματικότητα των οικονομικών ελέγχων συγκεκριμένη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας αλλά και για να καλυτερεύσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων αρμόδιων υπηρεσιών, των υπηρεσιών που αφορούν στην, στις οικονομικές πληροφορίες σε διασυνοριακό επίπεδο. Ευχαριστούμε η Έλγα Στίβενς επέστρεψε και έχετε το λόγο Έλγα. Ναι, δίκιο έχετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Μοσκοβισή, ως συνεισηγήτρια είναι αρμοδιότητά μου να προτείνω συγκεκριμένα μέτρα με προστιθέμενη αξία. Από το 2010 η Ευρωπαϊκή Ένωση ενταλλάσσε στοιχεία με τη ΣΥΠΑ σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Το σύστημα TFTP δεν περιλαμβάνει δεδομένα συναλλαγής σε ό,τι αφορά ε, μεταφοράς χρημάτων από υπουργό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πρόσβαση λοιπόν και γι' αυτό λοιπόν θέλουμε μια πρόσθετη ε, ανάλυση των δεδομένων αυτών. Το TFTS λοιπόν, το σύστημα αυτό. Καταλαβαίνω από τι Φάνηκε στη μελέτη φυκτότητα εντοπίστηκαν πολλά προβλήματα μεταξύ άλλων και το κόστο. Αλλά τέτοιο σύστημα θα χρειαζόταν Θα ήθελε η Επιτροπή λοιπόν να υπάρξει τέτοιο σύστημα και πώς θα λειτουργούσε το σύστημα αυτό. Μία εναλλακτική θα ήταν να υπάρξει κοινή διαμόρφωση του τμήματο οικονομικών πληροφορία προκειμένου να χρησιμοποιούν και ένα σύστημα το FIU-NET στα πλαίσια τη Europol και να ανταλλάσσουν πληροφορίε με άλλα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά το θέμα της ιδιωτικής σφαίρας, σε ό,τι αφορά τις οικονομικές μεταφορές. Είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα αυτό, αλλά χρειάζεται να υπάρχουν ευρωπαϊκά κριτήρια. Και ιδανικά, τι θα πρέπει να συμβεί για να υπάρξει καλύτερη συνεργασία στην καταπολίσμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Προσβλέπω στις ε, απαντήσεις σας, ε, Επιτροπή Μοσκοβισή. Ευχαριστώ. Merci, euh, Madame la Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο, επί... Επίτροπος. Είναι ερωτήματα που συμπίπτουν με σημεία στα οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση η πρότασή μας. Αναφέρεστε βέβαια σε αρμοδιότητες κάποιων συναδέλφων. Μόνο ένα σημείο που θέλω να σχολιάσω. Μιλάμε για τη δημιουργία ενός τμήματος οικονομικών πληροφοριών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δημιουργία ενός τέτοιου τμήματος είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα, την οποία θα πρέπει να αναλύσουμε επιπλέον, γιατί θα μπορούσε να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα στην καταπολέμηση της απάτης που, συγκρίνε, που άπτεται των τελωνίων και του ΦΠΑ. Στόχος μας είναι να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα συγκεκριμένα ζητήματα της απάτης των διασυνοριακών, των τελωνιακών μεταφορών και να μπορέσουμε να έχουμε ένα αρμόδιο νομικό όργανο που από κοινού μαζί με αυτό το τμήμα οικονομικών πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορεί να δρά από κοινού. Γι' αυτό και θα πρέπει να έχουμε μια οριζόντια προσέγγιση, κάτι το οποίο στηρίζει και η δική σας Επιτροπή. Και γι' αυτό και περιμένουμε τις δικές σας αντιδράσεις. Στα πλαίσια της οδηγίας για την καταπολέμηση του του ξεπλήματος του χρήματος που έρχεται από παράνομες δραστηριότητες. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό ένα τέτοιο τμήμα οικονομικών πληροφοριών. Εγώ προσωπικά λοιπόν με μεγάλη χαρά θα καλωσορίσω την δουλειά των συναδέλφων που αφορούν στη δημιουργία ενός τέτοιου τμήματος. Ευχαριστούμε πολύ. Η Άννα Γκομές λέει ότι το Κοινοβούλιο είχε προτείνει κάτι τέτοιο σχετικά με την οδηγία νούμερο 5 και ήταν το Συμβούλιο που ε, πλόκαρε την πρόταση αυτή. Ε, κύριε Πίτροπε, αγαπητέ Πιέρ, μπορείτε να απαντήσετε, λέει η Πρόεδρος. Στη Δανική γέφυρα για τέτοια θέματα. Ε, το έχω στη φύση μου, κάνω τη γέφυρα συνήθως. Και άλλωστε επειδή και προσωπικά μου είναι ιδιαίτερα προσφυλής αυτές οι ιδέες, θα κάνω την παρόν για να τις προωθήσω. Ε, νομίζω ότι από κοινού θα έχουμε καλύτερη και μεγαλύτερη δύναμη. Σίγουρα εν τη ενώσεις και είμαστε πολύ πιο στιβαροί και πολύ ε, πιο πιστικοί αν συνενώσουμε τις δυνάμεις μας. Θέλει άλλος κανείς το λόγο παρακαλώ γιατί έχουμε λίγα λεπτά ακόμη. Η Άννα ξέρω ότι έχει πολλά χαρτιά κατά το μανίκι της πολλούς άσους κρατάει και πολλές απορίες. Κύριε Επίτροπε, μερικές φορές ε, έχουμε περιπτώσεις όπου οι Αμερικανικές αρχές παρεμβαίνουν και ε, ζητούν κυρώσεις απέναντι σε ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικού οργανισμούς που εμπλέκονται σε νομοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητε, Είχαμε χαρακτηριστικό παράδειγμα της Μάλτας πρόσφατα, όπου μία τράπεζα που ε, εμείς είχαμε μάλιστα ε, προβληματιστεί πώς είναι δυνατόν να λάβει ο ιδιοκτήτης την ε, άδεια άσκηση τραπεζικών δραστηριοτήτων ενώ ε, έχει κατηγορηθεί στι Ηνωμένε Πολιτείε για παραβίαση του εμπάργου όπλων προς το Ιράν. Και έχουμε και την περίπτωση της Deutsche Bank και μιας μικρής ε, κυπριακής τράπεζας που έκλεισε ε, στο μεταξύ την FBME, αν δεν κάνω λάθο. Και εκεί βλέπουμε σαφείς διασυνδέσεις τραπεζών με εγκληματικέ δραστηριότητε, ενδεχομένω χρηματοδότηση τρομοκρατία και σίγουρα νομοποίηση εσόδων από παράνομε δραστηριότητε. Πώ ε, θα δραστηριοποιηθούμε ώστε να καταστήσουμε πιο αποτελεσματικές ε, τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές και πιο ευρηματικέ. Με ακριβώς αυτό είναι το ζητούμενο από όλους μας. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ε, διατάξεις για να ενισχύσουμε τα ευρωπαϊκά θεσμικά οργάνωση ευρωπαϊκούς φορείς χάρη στην καλή στο καλύτερο συντονισμό και συνεργασία και με ισχυρότερα νομοθετικά μέσα και μέτρα. Παρουσίασε ήδη τρεις νομοθετικές προτάσεις και με αύξηση των πόρων των αρμόδιων αρχών και φυσικά συνεργασία με τις Αμερικανικές αρχές. Και ας είμαστε σαφείς, ε, είναι θέματα που αρχίζουμε και τα πραγματευόμαστε μεταξύ μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά τα παγκόσμια θέματα θα πρέπει να εξετάζονται σε παγκόσμιους φορείς, στον νόσά για τα οικονομικά θέματα, στο G20 για την ανταλλαγή πληροφοριών και το καθεξής. Ευχαριστώ και η κυρία Μόνικα Χολμάγερ έχει μια νέα συμπληρωματική επερώτηση. Δεν μας είπατε τα περί χρυσού ε, διαμαντιών και άλλων τέτοιων πολύτιμων υλικών. Ε, και κατά δεύτερον, Στους οικονομικούς κύκλους τους οποίους συζητάτε, μιλάει κανείς για τα δισεκατομμύρια μουσουλμάνων, εύπορων από το Κατάρ, από τη Σαντική Αραβία, τα οποία χρηματοδοτούν ε, διάφορες οργανώσεις εδώ που είναι στα πρόσφυγα, θα έλεγα της ε, παρανομίας και προπαρασκευάζουν το έδαφος, προλιάνουν το έδαφος για ισλαμικές, ισλαμιστικές δραστηριότητες. Ε, γίνονται τίποτα συζητήσεις ε, για τα δισεκατομμύρια αυτά εύπορων οικογενειών, μουσουλμανικών οικογενειών που ενδεχομένως ε, χρηματοδοτούν και δραστηριότητες και Ισλαμικές ε, ροές και στα Βαλκάνια και μάλιστα σε πολύ μεγάλο βαθμό στη Βοσνία έχουν γίνει τέτοιες επενδύσεις δράστιες Συζητιέται το θέμα αυτό. Και τι μέτρα προτείνουν αν τυχόν ασχολούνται με το θέμα αυτό η οικονομική κύκλη σας. Κοιτάξτε, δεν μου έχει διαφύγει το γεγονό ότι δεν απάντησα 100% την απάντηση στην ερώτησή σας και δεν ε, είναι επειδή το ξέχασα, αλλά επειδή δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Είναι αλλονού αρμοδιότητα. Και εγώ αναγκαζόμαι να περιοριστώ στα δικά μου ζητήματα. Είναι θέματα στα οποία μπορεί να έχω τη δική μου προσωπική άποψη, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω σαν είναι δική μου αρμοδιότητα. Και να σας πω το οτιδήποτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Επίτροπε. Και νομίζω ότι στο σημείο αυτό απαντήθηκαν όλες οι ερωτήσεις των συναδέλφων. Και έχουμε την αίσθηση ότι υπάρχει μια πρόοδος. Έχουμε πλέον στη διάθεσή μας μια γκάμα εργαλείων τα οποία προετοιμάζονται ή έχουν ήδη υλοποιηθεί σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση τέτοιων επιθέσεων. Και χαιρόμαστε λοιπόν που έχουμε στη διάθεσή μας τα εργαλεία αυτά. Είναι τεχνικά φυσικά τα ζητήματα αυτά και μιλάμε από την άποψη αυτή. Γιατί πρέπει να εξηγούμε και στους πολίτες μας τι κάνουμε και τι πρέπει ακόμα να κάνουμε. Και όλες τις εργασίες με τις οποίες ασχολείστε, συνάδελφοι. Ο καθένας στον τομέα των αρμοδιοτήτων του. Και μάλιστα με αποτελεσματικότητα, αποφασιστικότητα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ που δεχτήκατε να έλθετε στην Επιτροπή μας και να ξέρετε ότι όλοι οι συνάδελφοι στην Επιτροπή μας θέλουν προς την ίδια κατεύθυνση να κινηθούμε για να πετύχουμε αποτελέσματα. Να προσθέσω και μια τελευταία κουβέντα, μου επιτρέπετε, κύριε ο Εγώ το κοινοβούλιο το εκτιμώ ιδιαίτερω και εκτιμώ τι εργασίε του. Δεν πιστεύω ότι πρόκειται για ακαδημαϊκέ ανταλλαγέ απόψεων ευγενικέ μόνο κουβέντε. Όχι, υπάρχει συγκεκριμένο πολιτικός αντικτύπο. Και έρχομαι εδώ για να απαντήσω στις ερωτήσει σας στον τομέα των αρμοδοτήτων μου, για να διαλευκάνω τι δράσει μου και θα ήθελα να μεταφέρω και ένα πολιτικό μήνυμα από δική σας πλευράς, γιατί η έκθεση σας θα έχει πολιτικό αντικτύπο, δεν έχω καμία αμφιβολία. Παρουσίασα λοιπόν τρία έργα, τρία projects τα οποία πιστεύω ιδιαίτερως και πιστεύω ότι είναι καινοτομικά και δείχνουν μία αποφασιστικότητα και θα έχουν αντικτύπο αρκεί να υλοποιηθούν και μια σε μια ειδική επιτροπή στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεωρώ ότι θα πρέπει να διαβιβάσετε το μήνυμα αυτό στους συναδέλφους σας το συντομότερο δυνατόν, όσο πιο γρήγορα, όσο πιο καλά. Το χωριό και εκεί. Αυτές οι τρεις προτάσεις λοιπόν που παρουσίασα. Κοιτάξτε, το ΦΠΑ είναι μεγάλο θέμα και είναι και πολύ περίπλοκο. Τα άλλα δύο όμως είναι και απλά και σαφή, ξεκάθαρα. Σε ό,τι αφορά τα πολιτισμικά αγαθά, δε, χάνουμε πραγματικά και δεν καταλαβαίνω τι περιμένουμε. Αν η έκθεσή σας, λοιπόν, μπορεί να μας βοηθήσει, να δώσει μια μικρή όθηση, ένα πρόξιμο, για να επιταχύνουμε τα πράγματα, εγώ θα είμαι αυτός που θα σας ευχαριστήσω για αυτά που κάνετε, αυτά που διαβιβάζετε προς τους συναδέλφους σας, γιατί το θέμα δεν είναι να κάτσουμε να αποφασίσουμε ποια είναι η αρμόδια επιτροπή και να τα συζητήσουμε. Το θέμα είναι πώς ε, θα καταφέρουμε να περάσουμε αυτή την πρόταση η οποία επαναλαμβάνω ότι είναι έτοιμη, απλή, ξεκάθαρη, ισορροπημένη και επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει να είμαστε γρήγοροι και ξεκάθαροι και τάχιστοι. Αυτό εκτιμούν οι πολίτες. Μάλιστα. Το λάβαμε το μήνυμα, λέει η Πρόεδρο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφοι. 23 Απριλίου η επόμενη συνεδρίαση τη Επιτροπή μα. 23 και 24 Απριλίου. Σα ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Σα ευχαριστώ και του συνεισηγητέ.